Ξεκινάμε τις εργασίες μας. Ε, να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με την χτεσινή συνάντηση των συντονιστών και θεωρώ ότι θα, έχετε, ε, ότι θα είναι εγκεκριμένα τα πρακτικά. Δεν έχω παρατηρήσει από τις προ... για τι προηγούμενε συνεδριάσει, αν δεν έχω παρατηρήσει από πλευρά σα. Ορίστηκαν δύο εισηγητέ για την έκθεση πρωτοβουλίας προβλήματα συνταγματικότητα μια ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστέ επέλεξαν έκαστο ε, μια την έκθεση αυτή, ε, αυτή την πρωτοβουλία που αξίζει τέσσερις πόντους. Δύο πόντους λοιπόν θα δώσουν οι σοσιαλιστές και δύο το ΕΛΚ. Ε, ε, όσον τώρα αφορά την γνωμοδότηση για την Επιτροπή Πολιτισμού για το πρόγραμμα Ευρώπη των Πολιτών, η συντάκτη συντάξη γνωμοδότησης θα οριστεί από την ομάδα των Πρασίνων για έναν πόντο. Για τη διαδικασία προπολογισμού 2013 ενδιαφέρονται οι σοσιαλιστές, αξίζει ένα πόντο και θα μας υποδείξουν τον εισηγητή για την έκθεση για την μετάφραση των ε, πρακτικών ε, της Ολομέλειας ε, θα ορίσει ε, εισηγητή η Άλντε. Που όμως εξέφρασε και μια επιφύλαξη για ανάκληση από το ενδιαφέροντος. Τώρα, για τις κοινέ προδιαγραφές για το διαδικασία ψηφοφορίας, ο εισηγητής θα οριστεί από το ΕΛΚ για έναν πόντο. Αποφασίστηκε επίσης να ζητήσουμε μια συγκριτική μελέτη από το τμήμα ε, θεματικής για τον δημοκρατικό έλεγχο και τη διαφάνεια και τις προθέσεις ψήφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα Εθνικά Κοινοβούλια των κρατών μελών. Θυμάστε ότι υπάρχει μια, ένα αίτημα για έκθεση πρωτοβουλίας από τον συνάδελφο Μέσερ Σμιτ, αλλά θεωρήθηκε ότι πρωτήτερα θα ήταν απαραίτητο να γνωρίζουμε τι συμβαίνει στα υπόλοιπα Εθνικά Κοινοβούλια, έτσι ώστε να έχουμε στοιχεία αξιολόγηση. Ε, επιβεβαιώθηκε ότι θα γίνουν επισκέψεις σε άλλες χώρες και η ημερομηνία είναι 18 και 19 Σεπτεμβρίου για τη Γαλλία, 20 και 21 Ιουνίου για τις ΗΠΑ, αν δοθεί η έγκριση, και 27 και 29 Νοεμβρίου για την Ιρλανδία. Προτάθηκε επίσης να αλλάξει η τακτική συνεδρίαση που είχε προγραμματιστεί 11, για τον Ιούλιο στις 11 και 12 Ιουλίου τελικά. Αυτές είναι οι αποφάσεις των συντονιστών Αν έχει κάποιους παρατηρήσεις να κάνει, ας τις κάνει. Δεν βλέπω να θέλει κανείς να πει τίποτα, οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε στην υπενθύμηση ότι η συνεδρίαση μαγνητοσκοπείται και μεταδίδεται στο ίντερνετ και τώρα έχουμε διάφορα να συζητήσουμε από ε, ε, τα, σημεία που πρέπει να συζητήσουμε και δεν είχαμε χρόνο να το μελετήσουμε. Χθες ήταν η έκθεση DAF για το πρωτόκολλο της ε, Δημοκρατίας της Τσεχίας. Θα έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσω με το σχέδιο Διεθνούς Συμφωνίας για την ενισχυμένη Οικονομική Ένωση και μετά να προχωρήσουμε στην ε, ψηφοφορία για την Τσεχία με κάποια εισαγωγικά λόγια του συναδέλφου Νταφ. Είναι εδώ ο συνάδελφος Γκουαλτιέρη που είναι ένας από τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου στην ομάδα εργασίας που είναι επιφορτισμένη με την εξέταση του σχεδίου Διεθνούς Συμφωνία και νομίζω πρέπει να του δώσω αμέσως το λόγο. Το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό το σχέδιο. Να δούμε αν έχουμε τα στοιχεία για μια πάνω κάτω οριστική πια αξιολόγηση. Παρακαλώ κύριε Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Η κατάσταση έχει ως εξή. Στις 19 Ιανουαρίου διανεμήθη στις 26 χώρες και στους παρατηρητές και στα όργανα το τέταρτο σχέδιο της Διεθνούς Συνθήκης το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο της συνεδρίασης που ε, διεξήχθη τη Δευτέρα το βράδυ Υπουργοί Οικονομικών, Οικονομίας των 26 συν την Κεντρική Τράπεζα, συν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επί τη βάση της έκβασης εκείνης της συνεδρίασης, ε, Έπρεπε να γίνει μια συνεδρίαση του ΣΕΡΠΑ αύριο που θα είχε ως έργο να τελειοποιήσει το σχέδιο το οποίο θα υποβάλαμε την επόμενη Δευτέρα στους επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων, ώστε αυτοί να ολοκληρώσουν τη συμφωνία και να μπορέσει έτσι να μεταφραστεί το κείμενο στις διάφορες γλώσσες για να το υπογράψει πρώτα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Έρινο ε, να το υπογράψουν 26 και μετά να πάει για την επικύρωση και όλη αυτή τη διαδικασία. Που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντό ενό έτου. Τώρα, όσον αφορά το περιεχόμενο, δεν θα επανέλθω στους λόγους ε, για τους οποίους έχει ασκήσει κριτική το Ευρωκοινοβούλιο για αυτή τη διεθνή συμφωνία. Δύο επικρίσεις, ε, μία θεσμικού τύπου, γιατί θεωρούμε ότι η Διεθνή Συμφωνία είναι, δεν είναι κατάλληλο ε, μέσο για να ενισχυθεί η διακυβέρνηση οικονομική της Ευρωζώνης και, αντίστοιχα, και αντίθετα μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό γιατί είναι μια συμφωνία που συνάπτεται εκτός του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και άρα θεωρήσαμε ότι θα ήταν καλύτερο να ενεργήσουμε μέσα στο πλαίσιο των συνθήκων ή αν υπάρχουν ε, ε, βάσιμοι λόγοι για αναθεώρηση της συνθήκης να κάνουμε μια αναθεώρηση. Πράγμα το οποίο δεν κατέστη δυνατό με, ε, λόγω του Βρετανικού βέτο, αλλά ε, να εξετάσουμε το κείμενο της ε, συμφωνίας με την εξαίρεση του, της διάσκεψης κορυφής του Euro Summit που με μια διεθνή συμφωνία δεν σημαίνει ότι γίνεται και ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Όλα τα άλλα που προβλέπει αυτή η συμφωνία θα μπορούσαν να γίνονται μέσω των κανονικών διαδικασιών που προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μόνο το Eurosummit δεν προβλέπεται. Το δεύτερο, η δεύτερη επίκριση, η διαφωνία μας είναι ότι αυτή η συμφωνία εστιάζει μόνο στο θέμα του προπολογισμού στην πειθαρχία του, του, την δημοσιονομική που θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη για την διατήρηση του ενιαίου νομίσματος, αλλά όχι επαρκή. Είναι απαραίτητη, αλλά όχι επαρκή η πειθαρχία. Υπάρχουν, χρειάζονται και άλλα μέτρα για να μπορέσουμε να εξέλθουμε τις κρίσεις ε, του δημόσιου χρέους. Παρ' όλα αυτά, το Ευρωκοινοβούλιο, όπως γνωρίζετε, ασχολήθηκε επικοδομητικά με τις διαπραγματεύσεις, βλέχθηκε ε, ε, στις διαπραγματεύσεις με στόχο να περιοριστεί η ζημιά σε νομικό επίπεδο για τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και για να προτείνουμε πιο αξιόλογες ε, διατάξεις που θα επιτρέψουν ε, την ε, ανάπτυξη και την αλληλεγγύη. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα για να... και είναι αυτή η στιγμή λεπτή για να κάνουμε τώρα απολογισμό του εργασία μας γιατί ακόμα βρισκόμαστε στις διαπραγματεύσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και αυτό κάναμε κάπως ε, επιφυλακτικό στις κρίσεις μου. Χωρίς όμως να σας κουράσω με τα διάφορα σκαμπανεβάσματα των διαπραγματεύσεων που έκανα το Κοινοβούλιο ε, να είναι πιο ε, ε, να έχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, κάποιες φορές να είναι πιο εκνευρισμένο άλλες φορές. Τώρα είμαι πιο αισιόδοξο ότι όλα, ορισμένα κομμάτια τις συμφωνίες αυτής που αφορούν την θεσμική διάσταση θα μπορέσουν να γίνουν τελικά δεκτά στο τελικό κείμενο αυτής της συνθήκης, όπως ε, πιο συγκεκριμένα τα εξή. Στο άρθρο 1 Φαίνεται να είναι πια και εκτιμένη η παρουσία μιας συμβολικής αναφοράς που ωστόσο είναι σημαντική στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση που δεν υπήρχε στο πρώτο σχέδιο. Στο δεύτερο άρθρο υπάρχει μια νέα επεξεργασία του διατύπωση μάλλον της τροπολογίας του Κοινοβουλίου για την ανάγκη εφαρμογής της συμφωνίας αυτής μέσω της δευτερογενούς ε, νομοθεσίας της Ένωσης όταν αυτό είναι δυνατό. Με αυτή την προστίκη, τη συμβιβαστική. Ε, στο τρίτο άρθρο θα πρέπει να πω ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να προκαλέσει και να ευνοήσει μια νέα διατύπωση πιο ευρεία που αν μη τι άλλο αφαίρεσε τον κίνδυνο μιας ε, αντίφασης με παραμέτρους ε, την μέτρηση του χρέους μέσα στο πλαίσιο του Διεθνού της Διεθνούς Συμφωνίας από αυτό που βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο της Ένωσης, δηλαδή το αναθεωρημένο στα, ε, σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και το εξαπλό νομοθετικό πακέτο. Από ό,τι φαίνεται η δική μας τροπολογία τώρα έγινε δεκτή. Θα έπρεπε να λέει medium term objective ως ποιοτική παράμετρο και ως ποσοτική παράμετρος παραμένει το 0,5 που εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ε, καλό για την ε, κοινοτική μέθοδο γιατί δεν έχει εισαχθεί στο εξαπλό νομοθετικό πακέτο ενώ υπάρχει εδώ αντί για το 0,1 αρθιωτικό μέσο πρόθεσμο χρέος. Ακόμα και αν υπάρχει δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση που θα το εντάσει και στη δευτερογενή νομοθεσία. Ίσως μάλιστα πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε, επικύρωσης ε, της συνθήκης αυτής εδώ. Όσον αφορά το άρθρο 4, το Κοινοβούλιο συνέβαλε στην πλήρη ευθυγράμμωση αυτού του άρθρου περί στην, με την κοινοτική νομοθεσία, ενίσχυσε ελαφρώς την διάσταση συντονισμού της, της έκδοσης τίτλων στο άρθρο 6, αν και δεν είναι απόλυτο συντονισμός, αλλά τουλάχιστον υπάρχει αυτή η βελτίωση που είναι πρόταση του Κοινοβουλίου. Για το άρθρο 9, αν αφαιρέθη η αναφορά στο σύμφωνο Europlus, Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αναφέρονται τα πλαίσια στα οποία θα πρέπει να ασκούνται οι πολιτικέ ανάπτυξη και στο άρθρο 10 και 11 γίνεται αναφορά στι κοινοτικέ διαδικασίε εφαρμογή των μέτρων για τη σύγκληση και την ανάπτυξη συγκεκριμένα άρθρο 136 για περί ενισχυμένης συνεργασίας. Και πάλι βρισκόμαστε στο πλαίσιο της διαδικασίας της Ένωσης και όχι εκτός. Το άρθρο 12, αυτό περί συμμετοχής, ε, παραμένει ανοιχτό όσον αφορά το θέμα των χωρών που έχουν εξαίρεση για το ευρώ. Ε, η Ένωση είναι υπέρ της πλήρου του σύνδεσης στις συνεδριάσεις του Euro Summit, ακόμα και αν στην αρχική, αρχικές πιο φιλόδοξες διατάξεις προτινόταν να θεωρηθεί το Euro Summit ένα διευρυμένο Eurogroup ώστε να μην ε, υπάρχει αυτή τη έννοια ενός νέου οργανισμού που δεν προβλέπεται από τις, ε, από τις συνθήκες και πλήρη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου πέρα από την διατύπωση που προβλέπει το 2.35 για το Ευρωσυμβούλιο που λέει μπορεί να προσκληθεί ε, για να μιλήσει. Αυτό είναι μια διατύπωση που λέει θα μπορούσε να δικαιολογήσει αυτή η διατύπωση. Ε, γιατί μιλάμε για ένα ξεχωριστό θεσμικό όργανο της Ένωσης, αλλά επειδή το Euro Summit θα είναι ένας άτυπος οργανισμός, δεν κατανοούμε γιατί θα πρέπει να προβλέπεται μόνο ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου να υπάρχει μια διαδικαστική, δηλαδή ε, ένας διαδικαστικός περιορισμός για τον τρόπο συμμετοχής του. Γι' αυτό θελήσαμε να, να διαγραφεί αυτή η αναφορά και να μιλήσουμε για συγκεκριμένη φυσιολογική πρόσκληση. Βέβαια την τελευταία λέξη θα την έχει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τέλος, όσον αφορά το άρθρο 13, είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αφορά τη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια και έχει περάσει η δική μας πρόταση για να τοποθετηθεί στο άρθρο 9 του πρώτου πρωτοκόλου. Η σημερινή διατύπωση αναφέρεται πιο συγκεκριμένα σε μια διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ε, Προπολογισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Επιτροπών ε, των αντίστοιχων μάλλον επιτροπών, δηλαδή η προϋπολογισμός και έκον του Ευρωκοινοβουλίου αλλά θεωρούμε ότι αργότερα θα μπορέσουμε να απλοποιήσουμε αυτή τη διατύπωση, αν υπάρξει τεχνική δυνατότητα. Πάντως αυτό που μετράει είναι η παραπομπή στο άρθρο 9 του πρώτου πρωτοκόλου που λέει ότι το Ευρωκοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια καθορίζουν μαζί από κοινού τον τρόπο συνεργασίας τους. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ότι ενώ στο άρθρο 14 φαίνεται ακόμα ανοιχτό, αν και φαίνεται να είναι 12 ο αριθμός των απαραίτητων υπογραφών για την έναρξη ισχύω της, Όσον αφορά και εδώ, σε σχέση με τους ε, αρχικούς εννέα, προσεγγίσαμε την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου και όσον αφορά το 16, το άρθρο 16, υπάρχει σε πιο αδύναμη μορφή δική μας τροπολογία για την ανάγκη να συμπεριληφθεί εντός 5 ετών η συνθήκη αυτή στο πρωτογενές ή δευτερογενές νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο δεν έγιναν δεκτές δυστυχώς οι δικές μας υποδείξεις με αναφορά στο θέμα του Ταμείου ε, σταθεροποίησης χρέους και πιο συγκεκριμένες ανα... δεσμεύσεις όσον αφορά την ανάπτυξη, ιδιαίτερα το ομόλογα έργου και ο φόρος πεπί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και όλα αυτά βεβαίω τα λέω με κάποια επιφύλαξη γιατί ακριβώ περιμένουμε τώρα τα συμπεράσματα. Δεν με μάλλον την ολοκλήρωση αυτών των διαπραγματεύσεων. Αν τα πράγματα εξελιχθούν λογικά, και αντικατοπτρίζονται τα σημεία αυτά που ενδιαφέρουν το Κοινοβουλίο και δεν αναφέρθηκα στα υπόλοιπα. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου ήταν καθοριστικός από την θεσμική πτυχή, γιατί περιορίσαμε τη ζημιά στο νομοθετικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και έτσι η συνθήκη αυτή ταιριάζει καλύτερα, αντιστοιχεί καλύτερα. Αν και υπάρχει εξισορρόπηση στις ουσιαστικές ε, πολιτικές, δυστυχώς ε, εκεί δεν μπορέσαμε να έχουμε τόσο μεγάλη επιτυχία. Εγώ εξακολουθώ να έχω έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά την, στερεότητα, την σταθερότητα της νομικής βάσης άρθρο, 1, ε, ε, άρθρο 8 συγγνώμη, και 8.1. Το 173 θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βάση για έναν ε, διατητικό ρόλο του, του, του, του δικαστηρίου δηλαδή όχι όπως προβλέπει το 263 και έχω ακόμα πιο έντονες επιφυλάξεις όσον αφορά τη δυνατότητα που προβλέπεται από το άρθρο 8.2 για να μπορεί το, το δικαστήριο να συνδυάζει κυρώσεις και ποινές ε, ε, ψυχαίοντας ε, την 2,73 με τη 2,60 χωρίς όμως καμία λογική νομική βάση. Όπως γνωρίζουμε όλοι δεν έχει καμία σχέση ε, αυτό του 2,60 με τον ε, διαιτητικό ρόλο του δικαστηρίου που προβλέπεται στο 2,73. Το ξέραμε εξ αρχής. Αυτό καθιστά αυτή τη συμφωνία όχι και πολύ σημαντική. Ε, στην ιστορία της ε, οικοδόμησης ε, μιας οικονομικής κυβέρνησης της Ευρώπης. Και επίσης δεν προβλέπεται υποχρέωση, υποχρέωση μάλλον του προπολογισμού και του golden rule, του χρυσού κανόνος, στο άρθρο 3 και κατά τη γνώμη μου αυτός ο μηχανισμός δεν θα είναι καθοριστικός στην επιβολή αυτής της συνταγματοποίησης του χρυσού κανόνα. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο είναι προτιμητέο αλλά δεν είναι δεσμευτικό. Περιμένουμε λοιπόν τα τελευταία κείμενα για να να κάνουμε την τελευταία μας αξιολόγηση που όπως είναι γνωστό δεν έχουμε καμιά υποχρέωση να δώσουμε ούτε γνωμοδότηση, συνένεση για μια συνθήκη που είναι μια διεθνή συνθήκη αλλά πώς τόσο. Ε, δεν μπορούμε να σιωπήσουμε εδώ. Και άρα η φύση της, της τελικής μας κρίσης θα εξαρτηθεί και από το πώς θα επιληθούν τα τελευταίοι γόρδιοι δεσμοί που έχουν παραμείνει. Γι' αυτό και επιφυλάσσομαι ώστε να εκφράσω τη γνώμη μου μετά από την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Δευτέρας. Σας ευχαριστώ. Πριν να ζητήσω από τον συνάδελφο Φερχώστα που, που να παρέμβει, αν θέλει, αν νομίζει πως είναι σκόπιμο. Εγώ έλεγα να το κάνω σε δεύτερο γύρο. Ώστε να μην ακούσετε δύο φορές τα ίδια πράγματα. Είμαστε τόσο ενωμένοι, τόσο συντονισμένοι. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πολύ ενωμένο. Αυτό θα πρέπει να το πω. Είχαμε πολύ ε, ενωμένη θέση σε αυτή την υπόθεση. Μάλιστα, ωραία, ευχαριστώ. Αν λοιπόν ο συνάδελφος Φερχόφστατ θέλει να λάβει το λόγο, θα το λάβει μετά από τις υπόλοιπες παρεμβάσεις. Πριν να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ταρκόφσκι, θέλω να χαιρετήσω τον συνάδελφο Βέμπερ, που είναι στην Επιτροπή μας νέος, ούτως υπήν. Πράγμα που ενισχύει πολύ το, το διανοητικό επίπεδο της Επιτροπής μας. Κύριε Ταρκόφσκι. Θα σας ε, πω το αγαπημένο μου εβραϊκό ανέκδοτο για την κατσίκα. Μπορεί και να το γνωρίζετε. Πηγαίνει ο Ίτσα στο Ραβίνο και λέει είναι η ζωή μου ένα χάλι, ε, έχω ένα πολύ μικρό σπίτι, μικρή κουζίνα, έχω έξι παιδιά, η γυναίκα μου συνέχεια γκρινιάζει, μένουν και οι πεθεροί μου και ο πατέρας μου, τι μπορώ να κάνω. Και του λέει ο Ραβίνος, αγόρασε μια κατσίκα. Γιατί λέει ο Ίτσα. Μη με ρωτάς, ε, πάρε την κατσίκα μόνο. Πάει μετά από μια βδομάδα ο, Ιτσακ στο, ο Ραφίνο και του λέει «Μα είναι τραγικά η κατάσταση, ε, πλέον τα κάνει και κουζί, κατσίκα στο σπίτι, μας έχει καταλερώσει, είναι βίωτη η κατάσταση». Όταν ε, λοιπόν ε, του λέω ο Ραβίνο διώξει την κατσίκα, πάει την επόμενη εβδομάδα και του λέει Α, τι ωραία, καταπληκτική ζωή μου κτλ. Αυτό μου θυμίζει την κατάσταση με το τρίτο σχέδιο και αυτό που έχουμε τώρα. very much relieved. Έχω ε, ε, ανακουφιστεί βλέποντας ότι αλλάζει η κατάσταση πλέον γιατί είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ιδίω σε σχέση με το τρίτο σχέδιο. Όπως είπε και ο διαπραγματεύτη, μας, βέβαια είναι πρόωρο να κρίνουμε τώρα την έκβαση, γιατί ακόμη είναι ρευστά τα πράγματα. Και σε ό,τι αφορά ε, τα θέλω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ελπίζουμε να γίνουν δεκτά, αλλά υπάρχουν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να τα προσέξουμε όταν θα αξιολογήσουμε το σύνολο του κειμένου. Πρώτα απ' όλα, η διατήρηση της κοινοτική μεθόδου, το ζήτημα της εφαρμογής. Αυτά έχουν τεθεί. Θέλουμε η εφαρμογή μέσω της δευτερογενούς νομοθεσίας κτλ. Όλα αυτά να ενισχυθούν στο κείμενο. Επίσης υπάρχει το ζήτημα της συμμετοχής των μελών της Ευρωζώνης, των μελλοντικών μελών της Ευρωζώνης στην όλη συζήτηση, ιδίω ό,τι αφορά τη συνεδριά της Ευρωζώνης. σε ό,τι αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων για την εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, θα πρέπει οι υποχρεώσει αυτέ να αναφέρονται πολύ ξεκάθαρα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Για το ρόλο επίσης του δικαστηρίου, ο Ρομπέρτο Καλκέρι μα είπε τα σχετικά, είναι ένα άλλο θέμα αυτό και υπάρχει και μια νέα ιδέα, δηλαδή η συμφωνία αυτή από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί, να δούμε ότι δεν θα πρέπει πλέον να αλλάξει χωρίς εμείς να μπορούμε να ελέγξουμε τη διαδικασία μετά από κάποιους μήνες. Ολοκληρώνοντας, ε, όπως και προείπα, μετά τις ανεπριγουμένου αλλαγές που πέστη το κείμενο από το δεύτερο σχέδιο στο τρίτο, δεν είναι περίεργο το ότι ανακουφιζόμαστε με την πρόοδο που βλέπουμε να έχει επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις και το ότι λαμβάνονται υπόψη κάποια από τα δικά μας αιτήματα, αλλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να περιμένουμε τον τελευταίο γύρο. Γιατί και πάλι μπορεί να έχουμε εκπλήξεις, όπως είχαμε πριν από δύο εβδομάδες στις 10 Ιανουαρίου συγκεκριμένα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Είπαμε στην αρχή ότι δεν μας ικανοποιεί η όλη διαδικασία. Και στόχος μας είναι να περιορίσουμε κατά τα δυνατόν τη ζημιά. Αλλά πρέπει να προσέχουμε και να μην προτρέχουμε. Στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό. Και θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Υπό την παρούσα του μορφή και είναι η τελευταία μου πρόταση, το κείμενο είναι πολύ καλό για να απορριφθεί ή για να το κατακρίνουμε. Ούτε και τόσο, αλλά είναι και κακό για να το επενέσει κανείς. Δηλαδή ούτε πολύ κακό, ούτε πολύ καλό. Ευχαριστώ. Grazie και τώρα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω ανέκδοτο να σας πω γιατί είναι πολύ πρωί ακόμα. να ευχαριστήσω τον Λουκαλτιχέρη, ε, του Μπλοκ και τον Φρεχόφστατ, που ήταν πολύ αποτελεσματική, Πολύ πιο αποτελεσματική από ό,τι θεωρούσα πιθανό στην αρχή του όλου εγχειρήματος. Κοιτώντας το τέταρτο σχέδιο, πρωτού δούμε το πέμπτο σχέδιο, μου έκανε εντύπωση ιδιαίτερα ο τίτλος του, που είναι ιδιαίτερα μεγάλος και αρκετά αν θέλετε, επιδεικτικός σε σχέση με τον προηγούμενο τίτλο. Νομίζω ότι για λόγους απλούστευσης και πιστότητα αν θέλετε ως προς τους πολίτες καλύτερο θα ήταν νομίζω να διευκρινιστεί λίγο ο τίτλος και να περιοριστεί στην έκτασή του για να αποτυπώνει την ουσία της συνθήκης και να μην την αποδυναμώνει ουσιαστικά. Θα το συζητήσουμε στην Ολομέλεια στις Βρυξέλλες την άλλη εβδομάδα. Και ενδεχομένως να προκύψει και ψήφισμα. Αν υπάρξει ψήφισμα, το σημαντικό είναι να μην λέει ότι αποτεχόμαστε, ότι συμφωνούμε τη συνθήκη αυτή, με τη συνθήκη αυτή. Μπορεί με να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για μια απαραίτητη ε, κίνηση στην παρούσα συγκυρία για την επίλυση της κρίσης. Αναγκαίο κακό. Αλλά να μην δώσουμε και ενδείξεις απόλυτης συμφωνίας από το Κοινοβούλιο. Ότι μην πούμε ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα το οποίο μα βρίσκει σύμφωνο απόλυτα προ την ουσία, του, την ουσία του. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί κατά την κατάρτιση του ψηφίσματο. Θα μπορούσαν να μας διαφωτίσουν οι συνάδελφοι σχετικά με το τι πιστεύουν κάποιες από τα συμβαλόμενα μέρη για τον απότερο στόχο της συνθήκης. Αυτό θα ήταν σκόπιμο ενδεχομένω. Και αυτό θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε ως Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Ντάφ. Το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφος Έφνερ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω καταρχάς ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι το Κοινοβούλιο με την ε, επιλεγμένη διαδικασία δεν έχει να πει ούτε τίποτα. Οι εκπρόσωποι του Ευρωπαίου πολίτη είναι καταδικασμένοι να μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα και να παρακολουθούν την κατάσταση. Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο μας έτρασε με ιδιαίτερη εξυπνάδα και αυτοί που έκαναν τις διαπραγματεύσεις και προσπάθησαν ένα αναγκαίο κακό κάπως να το βελτιώσουν, θα ήθελα να τους ε, ευχαριστήσω, γιατί νομίζω ότι προέκυψαν ε, ουσιαστικές ε, διαφορές. Το θέμα ποιο είναι, και θα πρέπει να συνεχίσει να είναι, να μην επιτρέψουμε γενικά στην Ευρώπη να παγιωθεί μία εξέλιξη όπου πολύ σημαντικές αρμοδιότητες για λήψη αποφάσεων θα λαμβάνονται εκτός των δημοκρατικά ελεγμένων οργάνων και επιτροπών και διαδικασιών. Δεν θέλουμε την Ευρώπη ενός νέου διακυβερνητισμού, όχι. Θέλουμε μια πιο δημοκρατική, πιο ενοποιημένη Ευρώπη. Και αυτό θα πρέπει να εκφραστεί και στη μεθοδολογία. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όλα αυτά ήταν πολύ χρήσιμα και ότι εν μέρη επιτεύχθη κάποια δέσμευση των αποφάσεων σε σχέση με αυτά που ισχύουν ήδη στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, αυτά που ψηφίστηκαν με το πακέτο των εξοδηγιών. Νομίζω λοιπόν ότι πέρα από αυτά τα οποία μπορούμε να διατυπώσουμε εδώ σήμερα, για μας ως Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το Κοινοβούλιο γενικά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, το βασικό έργο μας θα είναι στο μέλλον όλα αυτά που θα αναπτυχθούν ως παράλληλες δομές, αν θέλετε, ως doppelganger της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συγκεραστούν σε μία ενιαία Ευρώπη, σε μία ενιαία κοινωτική ευρωπαϊκή μέθοδο, με δημοκρατική βάση. Σε αυτά θα περιεριστώ σήμερα, γιατί αν θέλουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τις 10 τη συζήτηση, θα πρέπει όλοι κάπως να συντομεύσουμε. Eh, Μάλιστα, ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Γκερέρο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζετε ότι οι Ισπανοί, ή μάλλον οι περισσότεροι Ισπανοί, ε, Ερχόμαστε από μάλλον λέμε αστεία για τους Πορτογάλους ή για τους ε, Καταλανούς. Ε, δεν θα του πω εδώ τώρα του συναδέλφου Χάνζελ ε, τέτοιες πλάκες, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή η αντιζηλία μεταξύ μας υπάρχει εδώ και αιώνες. Να πω όμως ε, ότι Είναι, να πω όμως ότι είναι κάπως ε, παράξενη αυτή η πορεία που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από την πρώτη αυτή κρίση. Αυτές οι αλλαγές ε, γίνονται, συμβαίνουν όταν μετατρέπουμε τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε διαφορετικού τύπου προβλήματα. Ε, δηλαδή, λες και η διακυβερνητικότητα θα λύσει, τα, θα λύσει τα οικονομικά μας προβλήματα. Το Κοινοβούλιο είχε μια διαφορετική προοπτική και την ε, προοπτική που σχετίζεται με την ανάπτυξη, με τις πολιτικές επενδύσεων για να μπορέσει να φτάσει στην ανάπτυξη ανάπτυξη. Βλέπουμε τι αντιδράσει τι τελευταίε εβδομάδε των Ευρωπαίων ηγετών. Που ουσιαστικά δεν του ανησυχεί τόσο η λιτότητα, το ποσοστό, ε, πώ θα γίνει το ελλείμματο αποδεκτό. Αλλά αυτό που συζητούν είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει πιο ευέλικτο, πιο ελαστικό το χρονοδιάγραμμα τη μείωση του ελλείμματο για να μην υπάρξει εμπάθηση τη ύφεση που αυτή τη στιγμή βλέπουμε να υφίσταται όπως προτάθηκε από τα κράτη-μέλη, προτάθηκε ένα κανονιστικό εργαλείο, ρυθμιστικό εργαλείο, προσανατολισμένο αποκλειστικά και μόνο στην δημοσιονομική σταθερότητα. Και τώρα είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της δημιουργίας αυτού του εργαλείου, αυτού του μέσου. Τα περισσότερα πολιτικά μηνύματα ε, λένε ότι πρέπει ε, να την ξεχάσουμε αυτή την ε, δημοσιονομική σταθερότητα, την άκρο αυστηρή και να προσανατολιστούμε σε κάποιο άλλο είδος πολιτικών. Τι έγινε λοιπόν, τι έγινε, θα σας πω. Δεν επιλύσαμε το οικονομικό πρόβλημα. Άρα, η θέση του Κοινοβουλίου ήταν επισημάνει ότι αυτή η διακυβερνητική συμφωνία δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για να επιληθούν τα σημερινά οικονομικά προβλήματα στο δρόμο, όμως τελικά αυτό θέσαμε σε κίνδυνο την θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκή Ένωσης στρεφόμενοι σε διακυβερνητικούς μηχανισμούς και αποδυναμώνοντα τα σχετικά με την κοινοτική μέθοδο, ο ρόλος, ρόλο της Κομισιόν, ο ρόλο του Κοινοβουλίου. Όλα αυτά τα αποδυναμώσαμε. Αυτό το τελευταίο ζήτημα, κατά την άποψή μου, είναι και το ουσιώδες. Και εκεί πρέπει να επιμείνουμε κυρίως, γιατί θα μας δώσει και τη δυνατότητα να διαρθρώσουμε μια κοινή θέση, όλοι ενωμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, παρασπίζοντας όχι τη δική μας θέση, αλλά τη θεσμική δομή. Και καλό θα ήταν, αν είναι δυνατό αυτό, γιατί έχει γίνει σε προηγούμενες περιπτώσεις, καλό θα ήταν να συνεδριάσουμε, έστω και ανεπίσημα, πριν στην, την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ε, τεθεί το ζήτημα έγκρισης ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος δεν είμαι μεταξύ αυτών που θεωρούν ότι αυτό το σύμφωνο θα σώσει την Ευρώπη. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, στο Διεθνή Τύπο διαβάζοντα ε, διαπίστωσα ότι φαίνεται, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να έχει την ίδια θέση η Γερμανίδα Καγκελάριο, ε, που λέει ότι δεν θεωρεί πιθανό να μπορεί να σωθεί ούτε με αυτό το σύμφωνο, ούτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο η ελληνική οικονομία. Αυτά λέει τουλάχιστον ο διεθνής τύπος. Έχω ένα ερώτημα λοιπόν ε, προς ε, τους ε, εκπροσώπους μας από το Κοινοβούλιο. Σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση, τι αντιδράσεις βλέπετε, πώς βλέπετε τα πράγματα. Έρχεται ηγέτη, όχι μια οποιαδήποτε, αλλά ηγέτη, αν θέλει, τον χώρο τη Ευρωζώνη και κάνει μια τέτοια δήλωση. Πώ αυτό θα επηρεάσει την όλη διαδικασία, Grazie. Onorevole Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός κανόνας στην πολιτική. Να μην ρωτάς τίποτα αν δεν ξέρεις ήδη την απάντηση. Αν τηρούσα τον κανόνα δεν θα άνοιγα το στόμα μου, τέλος πάντων. Αν αυτή η συμφωνία έγινε χωρί ομόφωνη συμφωνία, άρα είναι μια ιδιωτική, ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, αν θέλετε, εκτό ε, πλαισίου Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ μπορεί λοιπόν να επιβληθεί ποτέ από τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Πώ θα είναι δεσμευτική θα είναι δεσμευτική. Αυτό είναι το ερώτημα. Βέβαια την απάντηση την ξέρω. ευχαριστώ και για τη συντομία κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και εγώ τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μάλλον τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πάρα πολύ ενεργητικά μας ε, ενημερώνουν και μας εκπροσωπούν. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί πολλά από όσα ήθελα να πω τα είπαν προλαλήσαντες. Δεν θέλω να επανέλθω στο θέμα της μεσονομικής ε, πειθαρχία, ε, αντικονομική σταθερότητα, ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη, ούτε θα επεκταθώ σε όλα τα θεσμικά σε όλες τις θεσμικές πτυχές που πάρα πολύ λεπτομεριακά ε, παρουσιάστηκαν, κοινοτική μέθοδος, ε, έναντι κτλ. Μας λείπει, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Το θέμα είναι να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη, η τελική πρόταση. Σε ένα συγκεκριμένο θέμα θέλω να ε, το, επεκταθώ. Η ενίσχυση της, της κοινοβουλευτικής διάστασης σε συνεργασία και με τα Εθνικά Κοινοβούλια, ενισχυμένη κοινοβουλευτική ε, εργασία που θα πρέπει να γίνει μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι ένα σημαντικό ε, στοιχείο, το τόνισαν ε, οι εκπρόσωποι μας. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, η Ένωση των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει ενισχυμένο έργο σε συντονισμό και συνεννόηση με τα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι καλό και μπορεί να δώσει η μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση σε αυτό το σχέδιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες τις επιτυχημένες σας προσπάθειες για την ενίσχυση του ρόλου όλων των κοινοβουλευτικών θεσμικών οργάνων φορέων. Ευχαριστώ. Και τώρα που είμαστε Έχουμε τρει διαπραγματευτέ. Ξέρουμε βεβαίω ότι έχουν εκφράσει ανέκαθεν ομόφωνη γνώμη, αλλά πιστεύω πω ο συνάδελφος Μπρόκ και ο συνάδελφος Φερχόφστατ ίσω θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν αυτή τη συζήτηση. Μπρόκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα και αυτό οφείλεται στο ότι ούτε εγώ ούτε το γραφείο μου φαίνεται ότι διαβάζουμε με προσοχή την ημερήσια διάταξη. Ο συνάδελφο Γκουαλτιέρη μα είπε προηγουμένω τα βασικά πράγματα, άρα δεν χρειάζεται να πει σε λεπτομέρειε. Ο κύριο Φερχόφσταϊτ και ο κύριο Γκουαλτιέρη και εγώ τα πηγαίνουμε αρκετά καλά και είμαι σίγουρος ότι αυτά που είπε ο κ. Γκουαλτιέρη με βρίσκουν σύμφωνο. Ουσιαστικά το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε την νομισματική πολιτική και την δημοσιονομική πολιτική της Ένωσης, αλλά να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και την κοινωτική μέθοδο. Αυτό μας φαίνεται ότι κάπως το πατήχαμε. Φυσικά το τελικό πόρισμα θα βγει Δευτέρα βράδυ μετά τη Σύνοδο. Αλλά φαίνεται ότι το πετύχαμε. θα γίνει η ρύθμιση με συναπόφαση με τους ε, κανόνες της συνθήκης. Και αυτό με αναφορά στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Και όπως είπε ο κ. Βαλτιέρ, δεν θα υπάρχουν διαφορετικά πρότυπα, θα πρέπει να ισχύει η κοινωτική μέθοδο Τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων φαίνεται ότι πλέον στη διατύπωση κατοχυρώνονται. Αν και φυσικά εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος μέχρι τελευταίας πτώσεως, μέχρι τελευταία στιγμής. σε ό,τι αφορά και τη συμμετοχή του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου στη Συμβούλιο. Όλοι οι συμβαλόμενοι εταίροι θα πρέπει με τον ίδιο τρόπο να μπορούν να συμμετέχουν στη σύμβαση και θα πρέπει να σε ό,τι αφορά τη, τη διαφορά που α, υπάρχει μεταξύ των κρατών και μη κρατών, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα πρέπει ε, να εξηγήσουμε όμως ε, και στα εθνικά κοινοβούλια γιατί επικυρώνονται τα όσα επικυρώνονται. Νομίζω λοιπόν ότι θα υπάρξει μεγάλη αντιπαράθεση στους κόλπους του Συμβουλίου. Η σύμβαση αυτή τρία πράγματα σημαίνει ουσιαστικά μόνο. Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει να κατοχυρηθεί ε, συνταγματικά στον εθνικό νόμο το φρένο στα χρέη. Κατά δεύτερον, ε, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρήση τη διαδικασία ελλείμματο. Αυτό περιλαμβάνεται στο πακέτο των έξι οδηγιών ουσιαστικά και για το άρθρο 126. Το τρίτο είναι ότι σε θέματα νομισματικής ένωσης θα πρέπει να συμμετέχει και το ΔΕΚ, το οποίο ρητά αναφέρεται στην, στην θήκη της Λισαβόνας. Μάλλον δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα στη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι πάντα προσέχαμε στις διαπραγματεύσεις ε, όλα τα υπόλοιπα να παραμείνουν στην κινητική μέθοδο και να μην ε, προκύψει διχασμός της Ευρώπης κατά τον τρόπο αυτό. Το ερώτημα για το ποια οικονομική πολιτική και ποια ισορροπία είναι η πιο σωστή ε, δεν ορίζεται στη συνθήκη, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αποτελεί μόνο ένας ακρογωνιαίο λίθος στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχίας. 3% για, τη συνολική, για την καινούργια χρέωση, 60% για τη συνολική χρέωση. Αυτή είναι, αυτά είναι τα μέτρα. Το θέμα είναι πώς θα τηρήσουμε σε βάθος χρόνου αυτόν τον κανόνα. Και μου δίνεται η εντύπωση πολλές φορές ότι πολλές φορές αμφισβητούμε και την τήρηση των δικών μας, των ίδιων μας των κανόνων που έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι. Και να ξέρουμε ότι αυτά τα δημοσιονομικά μέτρα από μόνο τους δεν πρόκειται να λύσουν την κρίση. Θεωρούμε όμως ότι ασφαλώς ε, ε, θα πρέπει να δοθούν οι παράγοντες για την επίλυση της κρίσης. Τα ορίσαμε τα στοιχεία αυτά πλέον στο κείμενο. Όλα αυτά περιλαμβάνονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό θεωρώ. Και υποθέτω ότι τη Δευτέρα θα προκύψουν και νέες προσεγγίσεις. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει να διαβάσουμε και την ομιλία της καγκελαρίου χτες στον Ταβός, όπου μιλήσαμε που μίλησα για μια νέα φάση στην ε, ανάπτυξη, για μια νέα διάσταση που θα δοθεί με την ε, σύνοδο αυτή και τη συνθήκη αυτή και θα πρέπει λοιπόν το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε αυτή τη νέα διαδικασία γιατί μόνο με οικονομίες θα πρόκειται να χρηματοδοτηθεί το έλλειμμα. Άρα λοιπόν με αυτό το πνεύμα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. ότι το θέμα των ευρωμολόγων δεν βρίσκει συμφωνία ούτε στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου, ούτε στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Είναι πολιτικό δεδομένο και σε ό,τι αφορά τον ε, φόρο επί των συναλλαγών. Να πω στον συνάδελφο Φόξ το εξή. Χαίρομαι που το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας προσπαθούμε να το πετύχουμε με τον τρόπο της Μεγάλης Βρετανίας, γιατί η Μεγάλη Βρετανία είπε ότι θα συμφωνήσει μόνο αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προβάλλει νομοθεσία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αυτά ήταν για την κρίση. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο μεγάλος τομέας να μείνει χωρίς ρύθμιση. Το ΑΕΠ όλων των χωρών όλου του κόσμου είναι 55 δισεκατομμύρια ευρώ. Και ο όγκος των χρημάτων που ρέει στον κόσμο χωρίς έλεγχο είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεκαπλάσιο, δεκαπλάσιο από την αξία όλων των κρατών σε όλο τον κόσμο. Άρα δεν μπορούμε να δεχόμαστε και στο μέλλον όλα αυτά τα χρήματα να κινούνται χωρίς ρύθμιση και να καταλύουν δημοκρατικές αρχές στα κράτη. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα... Δεν θα ήθελα να ακολουθήσουμε τη Βρετανική πρόταση για τη μη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Και όλα αυτά θα πρέπει να μείνουν και να γίνουν μέσω της κοινωτική μεθόδου. Με πλειοψηφικές αποφάσεις. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, έστω με ομοφωνία. Γι' αυτά θα πρέπει να, να προετοιμαστούμε. Πέρα από τη συνθήκη, λοιπόν, ε, θα πρέπει να προωθηθεί η νομοθεσία για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ευχαριστώ. Θέλετε, συνάδελφε Φερχόφστα, να πείτε κάτι ακόμα. Αν δεν το θεωρείτε πολύ τόσο απαραίτητο, όχι, αλλά αν θέλετε, έχετε το λόγο. Ε, Λίγα σχόλια, επιτρέψτε μου. Uh, Επειδή το ρώτησε ο κύριος Μέσσερ Σμιτ, έναν τρόπο για την ενίσχυση στο άρθρο 8, θα βρείτε τον τρόπο εφαρμογής της συνθήκης με το άρθρο 273 της συνθήκης, βάση του άρθρου 273 της συνθήκης. Πολύ ενδιαφέρον άρθρο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε 60 χρόνια το άρθρο 273, γιατί πρόκειται για ένα κράτος το οποίο αντιτίθεται σε ένα άλλο κράτος μέλος για θέματα που προκύπτουν και σχετίζονται με τη συνθήκη, που δεν είναι αντίθετα με τη συνθήκη, αλλά σχετίζονται με τη συνθήκη. Άρα, Εμείς τι προσπαθούμε να κάνουμε. Να δοθεί ένας ρόλος και στα κοινωτικά όργανα μέσω του άρθρου 273. Να μην πρόκειται μόνο για μία μάχη μεταξύ κρατών μελών, γιατί θεωρώ ότι είναι αδύνατον ένα κράτος μέλος να λάβει μία απόφαση στο κοινοβούλιο του να επιτεθεί σε ένα άλλο κράτος μέλος. Και για το λόγο λοιπόν αυτό, μετά από έτοιμά μας, ε, στο σχέδιο θα περιληφθεί σαφής ρόλος για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που καταρτίζει έκθεση σε περίπτωση που δεν τηρεί ένα κρατός μέλος κάποιες υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου 273. Όπως μας είπε ο Ρομπέρτο στην αρχή, τα πράγματα δεν ήταν ιδανικά, είναι μια αρχή και μόνο. Αλλά, εν πάση είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από την αρχική πρόταση. Πριν από κάποιες εβδομάδες. Άρα, Δεύτερη παρατηρήση, Πρόεδρε. Θα πρέπει να περιμένουμε το πολιτικό σχέδιο σήμερα. Έχουμε μετά συνάντηση σε ΕΠΑ αύριο, το Συμβούλιο τη Δευτέρα και μετά θα προκύψει το τελικό προϊόν, αν θέλετε, το τελικό αποτέλεσμα του εγχειρήματο. Και νομίζω ότι τότε θα πρέπει το Κοινοβούλιο να προβεί σε μια τελική αξιολόγηση, συνολική αξιολόγηση και να προετοιμάσει την άλλη εβδομάδα ένα σχετικό ψήφισμα, όπου καταρχάς θα εντοπίσουμε τα σημεία τα οποία τροποποιήθηκαν, κατά θετικό τρόπο, αλλά θα αναγνωρίσουμε και τις αδυναμίες της συνθήκης. Η συνθήκη λοιπόν αυτή πια τις αδυναμίες έχει, 99% ε, τίθεται στο δευτερογενές ε, δίκαιο. Επαναλαμβάνω αυτά που υπόθηκαν μετά, το τελευταίο, την τελευταία σύνοδο ΕΚΟΦΗΝ. 99% μέσω δευτερογενούς δικαίου. Και δεύτερη δυναμία της συνθήκης είναι ότι μιλάει μόνο για τη δημοσιονομική πειθαρχία και όχι για τα άλλα στοιχεία αλληλεγγύης. Νομίζω ότι τη δημοσιονομική την την αντιμετωπίσαμε. Έχουμε το six pack, το, το έχουμε τη συνθήκη, έχουμε τρία πλέον στοιχεία με τα οποία ενισχύουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία. Το πρόβλημα με την κρίση αυτή είναι ότι δεν κοιτάμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, το θέμα της αλληλεγγύης. Πώς θα μπορέσουμε να εξουδετερώσουμε, αν θέλετε, τα χρέη προκειμένου να πέσουν τα επιτόκια σε βιώσιμο επίπεδο. Γιατί α κοιτάξουμε την Ιταλία, για παράδειγμα. Μπορούμε να πούμε στον κύριο Μόντι να κάνει ό,τι θέλουμε και άλλε περικοπέ και άλλε μειώσει και άλλε ε, μειώσεις δαπάνε. δαπάνε. Αλλά τι θα κάνει άμα τα επιτόκια μένουν στο 6%. Δεν είναι βιώσιμο το επίπεδο αυτό. Άρα όλοι ξέρουμε ότι πέρα από τη δημοσιονομική πειθαρχία η οποία είναι απολύτω απαραίτητη θα πρέπει να υπάρξει και ένα σύστημα με το οποίο θα πέσουν τα επιτόκια για τις χώρες αυτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Στο Κοινοβούλιο, στις διαπραγματεύσεις, προασπιστήκαμε πάντα την ιδέα να τεθεί τουλάχιστον η ιδέα ενός Ταμείου Διάσωσης στην πρόταση. Ξέρετε ότι το Ταμείο Διάσωσης το έχουν προτείνει πέντε ε, γερμανοί οικονομολόγοι για να δημιουργηθεί ένα ταμείο 2,3 εκατομμυρίων ευρώ ώστε να μπουν όλα τα χρέη πάνω του 60% σε αυτό το ταμείο με ένα σχέδιο περικοπών σε όλη την Ευρώπη και μόνο οι χώρες αυτές που δεν θα συμμετέχουν στο ταμείο, που θα συμμετέχουν στο ταμείο διάσωσης δεν θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το ταμείο. Αυτό συνάδει με τη συνταγματική πραγματικότητα και με τη συνθήκη. Άρα δεν χρειάζεται αλλαγή ούτε συντάγματο ούτε τη συνθήκη. Άρα νομίζω ότι η πρόταση μια χαρά είναι, πολύ καλή. Τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα στο Κοινοβούλιο, να εξετάσουμε κατά πόσο είναι η συνθήκη μετά την ολοκλήρωσή της και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το επόμενο νομοθετικό πακέτο για να το πετύχουμε αυτό θεωρώ ότι ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσουμε με το Ταμείο Διάσωσης είναι να το συνδέσουμε με το πακέτο των δύο οδηγιών. Έχουμε το πακέτο των έξι οδηγιών που έχει τροποποιηθεί μετά από μακρές διαδικασίες και διαπραγματεύσεις και τώρα έχουμε το 2-PAC επιτάπητος στην Επιτροπή Οικονομικών. Είναι στην απόφαση, ε? Δεν είναι τα πράγματα όπως εδώ που μας καλούν να συμμετάσχουμε. Όχι, μιλάμε για συνομοθετική διαδικασία. Είναι λοιπόν καιρός να προετοιμάσουμε τη μάχη και το έταφος για το Ταμείο Διάσωσης. Να τεθεί ως ένα βασικό στοιχείο σε όλες τις συζητήσεις και σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για το ΤΟΥΠΑΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Νομίζω πως ε, τέλος θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε τους τρεις διαπραγματευτές μας, στον οποίο τις πλάτες ε, βασίζεται ολόκληρο το Κοινοβούλιο. Έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους, πολλά έχουν γίνει, είναι δύσκολη η κατάσταση. Ελπίζουμε πως θα διατηρηθούν αυτά τα επιτεύγματα και ότι θα πετύχουμε και κάτι ακόμα. Και τώρα να περάσουμε στη ψηφοφορία για την έκθεση για την τροποποίηση της πράξης περί της ή των μελών του Κοινοβουλίου την έκθεση ΤΑΦ και να καλωσορίσω τον ε, καθηγητή ε, Ζολάινεν για το οποίο η παρουσία υπογραμμίζει την σημασία αυτής της ψηφοφορίας που ήταν ήδη, έχει διατελέσει και πρόεδρος αυτής της Επιτροπής. Έχουμε όμως παραπάνω παρόντες από ότι ψήφους δικαιούται κάθε ε, ομάδα. Ο συντονιστή λοιπόν θα σας πει ποιος πρέπει να ψηφίσει και για τους σοσιαλιστές έχουμε έναν παραπανίσιο και για το ECR. Υπάρχει ένας παραπάνω. Να ψηφίσουν λοιπόν όσοι είναι μέσα στη σύσταση της Επιτροπής, σύνθεση της Επιτροπής. Για την πρώτη ψηφοφορία έχουμε να κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Eh? Allora, volevo ricordare... Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες. Να θυμίσω ότι η πρώτη ψηφοφορία αφορά την συμβαστική τροπολογία Ε σε μια προηγούμενη ε, λίστα ψηφοφορίας. Επειδή το ε καλύπτει την τροπολογία 15, αν εγκριθεί, είναι δίκαιο να ψηφίσουμε πρώτο τη 15 που αν εγκριθεί καλύπτει και την που καλύπτει το 1 και το 5. Ψηφίζουμε λοιπόν τη συμβιβαστική ε πρώτα. Παρακαλώ, όσοι είστε υπέρ να σηκώσετε τα χέρια σας. Bene, Εγκρίνεται γιατί είναι με προφανή συμπλειοψηφία. Να δούμε όμως αν υπάρχουν και κάποιοι που να είναι κατά. ένα είναι κατά. Αποχέ κανένας. Εγκρίνεται λοιπόν και καλύπτει όπω είπαμε την τροπολογία 1, 5 και 15. Περνάμε λοιπόν στην παράγραφο 1. Υπάρχουμε, έχουμε την τροπολογία 15 που ήδη καλύπθηκε. Έχουμε τώρα την τροπολογία 16. Ποιοι είναι η πέρα. Και κοντράριο. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στην τροπολογία 17. 18 και 18 και 19 διάφορες τροπολογίες ποιοι είναι υπέρ 5 και κοντράριο. κατά è ε, respinto απορρίπτεται περνάμε στην τροπολογία 20 Χέφνερ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε στην 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 22 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Παρακαλώ, σηκώστε τα χέρια σου, είστε υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική τροπολογία Α. Με μια προφορική τροπολογία. Κουαλτιέρη, θέλετε να μας εξηγήσετε. Ναι. Αντικατάσταση του καθορίζει με το προτείνει. Και έχει ζητηθεί και χωριστή ψηφοφορία για τα τμήματα. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα όπου υπάρχει η προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Και contrario. Κατά. Μόνο εγώ. Μόνο εγώ. Bene, è approvato. Ωραία, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Che riguarda la formula matematica, sì. E poi c'è la questione del resto del testo. Sulla formula matematica, chi è favorevole. Το δεύτερο τμήμα που αφορά το μαθηματικό τύπο. Ποιοι είναι υπέρ.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 Passiamo all'emendamento 24, è coperto dalle... 24 καλύπτεται από τη συμβιβαστική α, οπότε δεν την ψηφίζουμε. 27 δεν καταπίπτει γιατί άλλες τροπολογίες δεν εγκρίθηκαν, οπότε ψηφίζουμε την 27 Βίλαντ. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Σόλτς, ποιοι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26. Σέρεν, Σόντεργαρντ, υπέρ, κατά, αποχές,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 Περνάμε την... Ε, θα ψηφίσουμε πρώτα τη συμβαστική D. Ποιοι είναι περ. Κατά. Κανένας. Αποχές. Ομοφωνία. Η ψηφοφορία λοιπόν για την ε, ΔΕ συμπεριλαμβάνεται την τροπολογία 28, άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε επ' αυτής. Περνάμε στην τροπολογία J. Α, παρακαλώ κύριε Σιγητά. Ακούστε κύριε Πρόεδρε. Μετά από τις συνομιλίες που είχαμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα ήθελα να αποσύρω την προφορική συμβιβαστική πρόταση J Οπότε θα πρότεινα ανταυτή να υποστηρίξουμε την υπαριθμόν 29, ενώ είμαι αντίθετος με την τροπλή 30. Κατά αυτόν τον τρόπο καθορίζουμε και τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα. Σε τη λήψη απόφαση ε, για το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, κάτι το οποίο όλοι νομίζω προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να επιτύχουμε. Επομένως, επαναλαμβάνω, αποσύρω την και τροπολογία και ζητώ να στηρίξουμε την τροπολογία 29 του κ. Γκουαλτιέρη. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, συνάδελφε. Ντάφα, αποσύρεται λοιπόν η συμβαστική. J. ψηφίζουμε για την 29 του κ. Γκουαλτιέρη. Ποιοι είναι υπέρ, να σηκώσουν τα χέρια τους. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει έτσι η 30. le mettre comme, comme ajout. Caduc. Caduc. È caduc. Oui. Allora, emendamento 31. Περνάμε στην 31. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Β. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές έγκρινεται. Και καλύπτουμε έτσι και την 34. Πάμε στην 35. Κουαλτιέρη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36, Wieland, favorevoli. 36, υπέρ. Κατά. Τούτη. Αποχές, απορρίπτεται. Πάμε στη συμβιβαστική Ή. E. Ε, Ποιοι είναι υπέρ να σηκώσουν το χέρι του Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Και έτσι καλύπτονται οι τροπολογίες α, β και γ. ABC και η 42 και η 43. Paragrafo 11, 37. Chi è favorevole prima fa alzare la mano. Ψηφίζουμε για 37. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ΣΥ του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. δύο, τρεις είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται και καλύπτει τις 38 και 39 που δεν χρειάζεται να τις ψηφίσουμε. Και περνάμε στη συμβιβαστική D του εισηγητή, ποιοι είναι υπέρ. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Α, είναι ήδη γραμμένη εδώ. Μάλιστα. Ποιοι είναι υπέρ της συμβιβαστικής D. Να ψηφίσουμε, πείτε μου. Α, ψηφίσαμε ήδη. Ωραία. Α, σι-σί, grazie. Grazie, avevo dimenticato. Era già έχετε δίκιο, έχετε δίκιο, το έχουμε ψηφίσει ήδη πριν. Ε, το ξαναεγκρίναμε. Εντάξει, το ενισχύσαμε. 40, Ρανζέλ. Δεν θα την ψηφίσουμε αυτή, έχει καταπέσει γιατί υπερψηφίστηκε η συμβαστική D. Επίσης ε, ε, καλύπτεται η τροπολογία 1 την οποία είχαμε ψηφίσει την συμβαστική ε. Πάμε στην τροπολογία 2 Γουαλτιέρη. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Γουαλτιέρη. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική F του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καλύπτεται 4. Η 5 ήδη έχει καλυφθεί από την άλλη συμβαστική ε, την οποία ψηφίσαμε προηγουμένω και ψηφίζουμε την 6 στο εκτιμώντα 1 του Κουαλτιέρη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται. Είμαστε στην τροπολογία 7, Κουαλτιέρη. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική G, υπέρ. Κοντράρι. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 έχει καλυφθεί. Πάμε στην συμβιβαστική H. Ποιοι είναι υπέρ. Και κοντράριο. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Όχι, θα το ψηφίσουμε χωριστά. 10 λοιπόν υπέρ. Μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί τη 10 και την 11 γιατί είναι ταυτόσιμες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 12. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 13 και 14 από κοινού είναι ταυτόσιμες και άρα μπορούμε να ψηφίσουμε μόνο μία φορά 13 και 14 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται και περνάμε έτσι στην τροπολογία 43 ανακαλύπτεται. Ah sì sì, chiedo scusa. No. Sì, il protocollo 7 è già stato. Benissimo. Allora siamo al voto finale. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. 15, 16, 17. 17. 17 contrari. Cata. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contrari. Astenzione. Astenzione, nessuno perché siamo Astenzione. Astenzione. Una. Κατά μετρήσαμε. Αποχές ποιος είναι, ποιος απέ. Α, είναι κατά. Είστε κατά. Mm. Allora, era, allora, allora era nel, nel contrario 17 contro 7 17 contro 7 in sostanza 17 υπέρ 7 κατά λοιπόν αυτά εγκρίνεται λοιπόν κύριε Ντάφ ο κόπος σας τουλάχιστον ανταμείφθηκε πιο δύσκολο θα είναι στην Ολομέλεια μπορούμε να προχωρήσουμε με την ψηφοφορία για την άλλη έκθεση, πάλι του κυρίου Ντάφ. Il protocollo relativo alla Repubblica Ceca Λοιπόν, η επόμενη είναι το πρωτόκολλο για την ε, Δημοκρατία της Τσεχίας. Κύριε Ντάφ, σύντομα όμως. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε. Απλά δεν καταφέραμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες ό,τι αφορά το πρωτόκολλο για την ε, Τσεχία εχθές. Θα ήθελα λοιπόν ε, πολύ σύντομα να σας επενθυμίσω Γιατί ο συγκεκριτής σας είναι αντίθετος με την εξέταση του αιτήματο αυτού της τσεχικής δημοκρατίας της πρώην κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Κατά την άποψή μου, το υπαριθμόν 30 πρωτόκολλο, στο οποίο θέλουν να επιδιώκουν να ε, προσχωρήσουν οι Τσέχοι, είναι από την αρχή, για ένα, ε, είναι από την αρχή ένα εργαλείο το οποίο επινόησε ο κύριος Μπλερ για να πείσει τότε τη Βουλή των Κοινοτήτων, γιατί στη Βρετανία υπήρχε το opt-out της ε, Βρετανίας από το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εξ τότε αποφάσισε και αποφασίστηκε και από την ομολογία, μάλλον επιβεβαιώθηκε αυτό, ότι Είχε λάθος ο κύριος Μπλερ. Δεν υπάρχει αυτό το opt δεν είναι σωστό. Και από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη του πρωτοκόλου ουσιαστικά είναι περιττή. Είναι περιττό το πρωτόκολλο αυτό, για να μην πω ότι δημιουργεί και ανασφάλεια ε, δικαίου και πολιτική σύγχυση. Το Κοινοβούλιο ποτέ δεν το υποστήριξε. Ούτε και το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Χθε ε, από την Προεδρία ο κ. Βάμεν μας είπε ότι το Συμβούλιο ουσιαστικά πρέπει να κάνει το καθήκον του και να στηρίξει το αίτημα αυτό της ε, τσεχικής κυβέρνησης. Διότι αυτή είναι η δουλειά του. Ε, αυτή είναι η αρμοδιότητά του. Το κοινοβούλιο μας όμως λειτουργεί διαφορετικά. Μας δείτε λοιπόν να συντάξουμε μια γνωμοδότηση, να δώσουμε την άποψή μας. Η δική μου άποψη είναι αρνητική. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να απορρίψουμε όλες τις τροπολογίες. Θα ζητούσα να προστατεύσουμε την ακαιρεότητα αλλά και την αξιοπιστία του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. Αν θέλει κάποιο να παρέμβει, μπορεί, γιατί το σημείο αυτό ήταν προ συζήτηση χτε το βράδυ. Παρακαλώ, κύριε Μπρόνς. Όχι, κύριο Μπόργο. Prego. Prego. za já se já dobře nerozuměla eh, eh, Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Ε, απλώς θέλω να μιλήσω για αυτά τα δικαιώματα. Ε, στα δύο σώματα του Κοινοβουλίου ψηφίσαμε το 2009 τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν θέσαμε καμία προπόθεση, κανέναν όρο. Υπάρχουν ε, δύο ζητήματα σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, τη συνθήκη της Λισαβόνας έπρεπε να είναι συμβατή με το τσεχικό σύνταγμα. Η τσεχική δημοκρατία Ξεκίνησε κάποιε διαδικασίε πράγματι, ε, μέσω του Προέδρου για προσχώρησή τη στο πρωτόκολλο υπαριθμό 30. Αυτό το πρωτόκολλο είναι απόλυτα συμβατό με το Σύνταγμά μας. Από την άλλη πλευρά, το ζήτημα δεν έχει ρυθμιστεί. Δηλαδή, ε, ναι, η Τσεχική Δημοκρατία στήριξε, επικύρωσε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το πρωτόκολλο 30. Εμείς ζητούμε ειδική εντολή. Η Άνω Βουλή, η Γερουσία δηλαδή, στο Τσεχικό Κοινοβούλιο, έθεσε ένα αμφιβόλο το σκόπ, τη συνταγματικότητα του πρωτοκόλλου 30 σε σχέση με το χάρτη θεμελιών δικαιωμάτων και υποστηρίζει ότι θα έχει ε, μια ε, επίπτωση, έναν αντίκτυπο. Αυτό το πρωτόκολλο που υπερβαίνει ουσιαστικά το πεδίο του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Έχουμε αναλύσεις από εμπειρογνώμονες, ιδίως ε, από το τμήμα της νομικής του Πανεπιστημίου μας έναν καθηγητή που είχε πει ήδη από το 2009 ότι δεν μπορεί το πρωτόκολλο αυτό να θεωρειται οπτά, ότι ξέρεις από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως ερμηνεύεται Πάντως θα έχει σημαντική νομική επίπτωση, αντίκτυπο αυτό το πρωτόκολλο. Μάλιστα θα έχει και κάποιες ε, πολύ σημαντικές συνταγματικού χαρακτήρα συνέπειες. Και πρέπει να δούμε και τι ε, θα συμβεί και με τις εξουσίες του δικαστηρίου δυνάμει αυτού του πρωτοκόλου που θα διευρυνθούν. ουσιαστικά θα περιοριστούν κατά την άποψή μας τα κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών της Τσεχικής Δημοκρατίας με την εφαρμογή του, του πρωτοκόλου και θα υπάρξει και ασάφεια νομική. Επομένως, σας ε, παρακαλώ και εγώ να στηρίξετε τον κύριο Νταφ και να μην δοθεί συνέχεια στην υπόθεση αυτή. Bene, grazie. Adesso ha chiesto la parola l'onorevole σας ευχαριστώ. Έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Σεφλίν. Θα είμαι σύντομο, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ξεκάθαρο παράδειγμα της απόκλησης που υπάρχει μεταξύ πολιτικής και νόμου, δικαίου. Ποια είναι η πολιτική διάσταση. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έγινε μια, εδόθη μια υπόσχεση. Για όποιο λόγο και αν έγινε αυτό, οι ιστορικοί θα το αποφασίσουν. Ο κύριος Νταφ πάρα πολύ καλά τα είπε για αυτή την συμφωνία τελικά που είχε γίνει τότε. Αλλά έγινε υπόσχεση, δόθηκε και θα πρέπει να την τιμήσουν. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Πράγματι δεν είναι ξεκάθαρο. Συμφωνώ, υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ της Άνω και Κάτω Βουλής. Ίσως κάποιο θα έπρεπε να το χρησιμοποιήσει αυτό σε επιχείρημα υποστηρίζοντας ότι το κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει μόνο ένα σώμα και όχι δύο. Ε, τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή ότι ε, η πολιτική δέσμευση που έχει αναλυφθεί πρέπει να τηρηθεί. Αυτό είναι το θέμα κατά την άποψή μου. Κύριε Μπρόνς, μάλιστα. Ο κύριος Ντάφ αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Τόνι Μπλερ. Φαντάζομαι ότι αναφέρθηκε σε, αυτό, σε αυτές τις δηλώσεις λέγοντας ότι δεν υπήρχε βλάβη για το, από την, ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω, τόσο προκατηλημένος ήταν και ποιος τον ε, παρέσυρε τόσο πολύ. Στην ουσία θέλουν να μας αναγκάσουν να υπογράψουμε την ε, στη Συμφωνία της Λισαβόνας. Όχι μόνο λοιπόν στερήθηκε το εκλογικό σώμα της Βρετανία ενός ε, δημοψηφίσματος, αλλά ε, στερήθηκε και στη... Ε, το ίδιο το, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, η Βουλή των Κοινοτήτων. Δεν θέλω να προτείνω βεβαίω ότι ο κύριος Νταφ έχει δώσει σαφή λογαριασμό. Αυτό που έκανε είναι να δώσει ένα σαφή λογαριασμό σύγχυσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, η κατάσταση που περιγράφεται είναι περίπλοκη και αντιφατική και μας δώσατε πολύ σαφή λογαριασμό για όλα αυτά. Αλλά δεν καταφέρατε να τα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα για μας. Μου θυμίζει κάπως εκείνο το κομμάτι στα ταξίδια του Γκάλιβερ, όπου ο Γκάλιβερ μιλούσε για τις θρησκευτικέ διαφορές στην, στην Αγγλία και έλεγε ότι ήταν οι ε, λίλιπούτη και οι άλλοι, αλλά βέβαια αυτό δεν έχει και ότι όλοι τσακώνονταν για το πού θα πάνε, αλλά τελικά δεν είχε και πολύ σημασία και τελικά όλοι το ίδιο τέλος θα έχουμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο βέβαια συμβαίνει το αντίθετο, ότι ο ένας θέλει να μην επιτρέψει την ε, περάση νομοθεσία, ο άλλος θέλει να εφαρμοστεί σωστή νομοθεσία, αλλά τελικά και οι δυο καταλήγουν στην, ίδιο, στην ίδιο παρονομαστή, δηλαδή ότι το opt-out είναι καλύτερο. Θέλει ο κύριος Ντάφ να απαντήσει και μετά να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Εν συντομία, σε απάντηση στον κύριο Μπρόνς, θα ήθελα να συστήνσω στον κύριο Μπλερ, επειδή είχα το προνόμιο να προσπαθήσω να τον συμβουλέψω για το θέμα αυτό ως παλαιό μέλος της συνέλευσης που κατήρτισε το χάρτη. Η συμβουλή μου όμως δεν έγινε αποδεκτή και τελικά καταλήξαμε σε αυτά τα χάλια. Δεν νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μαζέψουμε τα χάλια αυτά τώρα. Bene, passiamo allora alla, ai voti. Come sapete i documenti sono due, anche se il contenuto è lo stesso. Il primo riguarda proprio il merito, il secondo riguarda la decisione della... Λοιπόν, πάντως πρέπει να ψηφίσουμε και Τώρα, εμείς θέλουμε να ζητήσουμε λοιπόν ε, συνέλευση. Λοιπόν, περνάμε στην, ψηφοφορία για το πρώτο Η Πρώτη τροπολογία είναι η, παρα... η τροπολογία 3 που υπέβαλε ο Μέντες Δεβίγκο και τώρα στηρίζει ο συνάδελφος Σόφλίν. Ποιοι είναι υπέρ.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 Τροπολογία 1. Μέσερ Σμιτ. Υπέρ. Κοντράρι. Κατά. Ε, come stiamo? Contrari. Non è Κατά. Τροπολογία 2. Τώρα. Στην ε, τελική σκέψη M. Υπέρ. Contrari. Κατά. Ε, respinto. Απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν στην τελική ψηφοφορία. Για ολόκληρη την έκθεση. Ποιοι είναι υπέρ, να σηκώσουν τα χέρια τους.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 φαίνεται να είναι ότι το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να γνωμοδοτήσει στο... προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό αποτελεί την τελική μας θέση. Η δεύτερη απόφαση η οποία θα πρέπει να λάβουμε για την συνέλευση

Μετά από διαβούλευση εδώ με τη γραμματεία φαίνεται να είναι περίπλοκα τα πράγματα, γιατί το κοινοβούλιο έχει την υποχρέωση να συντάξει γνωμοδότηση. Δεν είναι δηλαδή ότι κάνουμε το καθήκον μα δεν δώσαμε τη γνωμοδότησή μα, όμω το Συμβούλιο μπορεί ούτως ή άλλως να προχωρήσει. Μήπως είμαστε υποχρεωμένοι. Άρα πρέπει αυτό και από την αρχή να ξεκινήσουμε. Δεν έκλεισε το ζήτημα. Μάλιστα. Όχι, δεν έκλεισε το θέμα. Δεν ήμασταν σε θέση να εκφράσουμε την ε, γνωμοδότηση που είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, τώρα ε, υπάρχει και το θέμα της σκοπιμότητας. Και ρωτώ τη συμβουλή του κυρίου Νταφ αν πρέπει να ψηφίσουμε για το άλλο θέμα, αν είναι σκόπιμο ή να όχι να κάνουμε συνέλευση. Εγώ νομίζω πως ε, ούτως ή άλλως είναι σκόπιμο, αλλά ε, να ψηφίσουμε και για το δεύτερο θέμα. Συνάδελφε Εντάφε, τι νομίζετε. Νομίζω ότι επί της ουσίας της γνωμοδότησης οι συντονιστέ μπορεί να συνεχίσουν τη συζήτηση για το κατά πόσο θα κάνουμε κάτι διαφορετικό ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχω την αίσθηση ότι σήμερα δεν είναι κατάλληλη η ημέρα να προχωρήσουμε για το θέμα αυτό. Ούτε να αποφασίσουμε για το κατά πόσον θα υπάρξει ή όχι συνέλευση. Θα προτιμούσα να ανασταλεί η διαδικασία. Αυτή είναι η γνώμη του εισηγητή. Οι υπόλοιποι Συμφωνείτε. Αν συμφωνείτε μπορούμε να δεχτούμε αυτή την ιδέα της αναστολής. Ωραία λοιπόν. Το αποφασίζουμε έτσι. Και τελειώσαμε τη διαδικασία ψηφοφοριών. Πάμε λοιπόν στο σημείο 15. Allora, eh, su richiesta della Commissione europea, κατόπιν ετήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και κατόπιν προτάσεως ε, του δικού μας, Χέφνερ, που είναι εισηγητής για τη γνωμοδότησή μας προς την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, η εκπρόσωπος ε, της Επιτροπής, η κυρία Μπέρναρτς, έχει προσκληθεί στη σημερινή μας συνεδρίαση για να μας ε, παρουσιάσει την πρόταση της Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών το 2013. Αν λοιπόν τα καταφέρναμε κάπως να κάνουμε ησυχία... Se riusciamo a fare le conversazioni fuori Αν καταφέρναμε να κάνουμε και τις συζητήσεις μας. Θα παρακαλούσα την κυρία Μπέρναρτ να μας παρουσιάσει αυτή την πρόταση της Κομισιόν για το, έτος, το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών. Παρακαλώ. Thank you, Chair, for... Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που με καλέσατε να παρουσιάσω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ε, απόφαση για το Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη το 2013. Κυρίες και κύριοι, θα θυμάστε ότι το Δεκέμβριο του 2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διοργανώσει το έτος αυτό για να δώσει μια ορμή, αν θέλετε, για την πρωτοβουλία των πολιτών και για να ενημερώσει τους πολίτες για τα δικαιώματά τους. Το Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη το 2013 θα λάβει χώρα σε ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο, ένα έτος πριν τις ευρωεκλογές του 2014 και επίσης στην 20η επέτειο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας την οποία εισήγαγε η συνθήκη του Μάστριχτ. Αλλά ξέρουμε ότι διανύουμε και δύσκολου καιρού οικονομική και δημοσιονομική κρίση και χρειάζονται πιο πολλέ προσπάθειε παραποτέ για να ενθαρρυνθεί ο κόσμο να συμμετάσχει ενεργά στο ευρωπαϊκό έργο και για να εξηγήσουμε καλύτερα τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρωπαϊκό έτος βασίζεται σε τέσσερις βασικές ιδέε. Οι Ευρωπαίοι διαρκώς συνδέουν την ευρωπαϊκή ηθαγένεια με την ελευθερία κινητικότητα για σπουδές, για επιχειρήσεις και το καθεξής. Θέλουμε το ευρωπαϊκό έτος να επισημάνουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στους πολίτες και τα ενδεχόμενα ωφέλη. Η συζήτηση θα ξεπεράσει τα δικαιώματα της ελεύθερης κίνησης. Θα περιλαμβάνει τα δικαιώματα εκλογής, ε, της ε, πρωτοβουλίες των πολιτών, δικαιώματα υποβολής ε, αιτήσεων και θα δώσει συγκεκριμένο μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια και απάντηση σε προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολιτής καθημερινά. Το... Η αναφορά σε δικαιώματα που απασχολούν τον πολίτη θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω συζητήσει. Και νομίζω ότι το ευρωπαϊκό έτο θα συμβάλλει στην ανάκτηση τη εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε σήμερα σε εποχές κρίσης ε, επιπλέον δυνατότητες στον Ευρωπαίο πολίτη. Είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ, προκειμένου να λαμβάνουν αποφάσεις για την ίδια τους τη ζωή και που θα βοηθήσουν την ε, δημοκρατική ζωή το δημοκρατικό βίο σε όλα τα επίπεδα και υπάρχει ε, άμεση σχέση μεταξύ των πολιτικών δικαιωμάτων της, ε, και της συμμετοχής στην πολιτική ζωή. Θα πρέπει να συνεχιστεί ένας ευρύς διάλογος μετά από όσα έχουν ξεκινήσει το 2010. Η αύξηση λοιπόν αυτής της ευαισθητοποίησης δεν μπορούν να αποτελέσουν αυτό σκόπο. Το 2013 θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματο του ανήκει και του αισθήματο της ευθύνης ε, και τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτουν και συγκεκριμένα δικαιώματα και ευκαιρίε χάρη σε μια ευρεία προσέγγιση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας Καταρχάς, ε, το έτος αυτό θα αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία για να καταδειχτεί ότι οι πολίτες είναι στον πυρήνα της πολιτικής ατζέντα και να εξηγηθεί τι σημαίνει ακριβώς η πολιτική ηθαγένεια. Και αυτό θα δώσει την ε, δυνατότητα να εξηγηθούν βασικά ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες θα πρέπει να είναι ένα έτος για τους πολίτες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τα άλλα θεσμικά όργανα, με το Κοινοβούλιο, με την Κοινωνία των Πολιτών, με τις εθνικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η προσέγγιση αυτή θα πολλαπλασιάσει σημαντικά τα ενδεχόμενα αποτελέσματα και τον πολιτικό αντίκτυπο λοιπόν του έτους. Θα ήθελα να τονίσω με σαφήνεια ότι το ευρωπαϊκό έτος ε, ε, συμπεριλαμβάνει και την χρήση διαφορετικών μέσων και εργαλείων. Θα δημιουργήσει μία κληρονομία προωθώντας όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νομοθεσία, έχει πρόγραμμα χρηματοδότησης, έχει διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε όμως μέσα από τα μάτια του πολίτη, κατανοώντας τις προσδοκίες του πολίτη. Ξέρω ότι κάποιοι εξήμων ανησυχείτε σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Έτους για τον πολίτη. Δύο θέματα εδώ έχουν σημασία. Πρόκειται για ένα πολιτικό μήνυμα σε εποχές λιτότητας. Ο κόσμος που βλέπει τους μισθούς του να μειώνεται μπορεί να ανησυχήσει όταν βλέπει ότι για επικοινωνιακά μέσα χρησιμοποιούνται τεράστιοι προϋπολογισμοί. Από την άλλη, το ευρωπαϊκό έτος αυτό δεν αποτελεί μια απλή εκστρατεία ενημέρωσης. Ε, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με πολλούς ε, φορείς που μπορούν να αναφερθούν σε θέματα που απασχόλουν τον Ευρωπαίο πολίτη. Πολλά μέσα θα χρησιμοποιηθούν και μάλιστα τα πλέον κατάλληλα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του πολίτη. Ως εκ τούτου το Ευρωπαϊκό Έτος θα αποτελέσει μια πρακτική απόδειξη του τι σημαίνει να βάζουμε τον πολίτη στο κέντρο της ευρωπαϊκής ε, δράσης. Θα ξεκινήσει μια κεντρικά διοργανωμένη εκστρατεία ενημέρωσης. Σκοπός μας δεν είναι μόνο να ενημερωθεί ο πολίτης για τα δικαιώματά του, αλλά να λάβουμε και ένα feedback, μια απάντηση αν θέλετε για το τι θα διευκολύνει τον πολίτη στην καθημερινή του δράση και στην πολιτική του δράση θα υπάρξει και μια ιστοσελίδα, θα υπάρχει ένα εργαλείο, αν θέλετε, ένα κυβότιο με εργαλεία επικοινωνιακά και διάφορα τέτοια ε, μέσα σε εθνικό επίπεδο. Η σχετική έκθεση θα αποτελέσει και επίσης μια βάση για συζήτηση και θα μας δώσει συγκεκριμένα αποτελέσματα στο τέλη του χρόνου. Θα διοργανωθούν αρκετά, αρκετές εκδηλώσεις με την κοινωνία των πολιτών, με τις δύο προεδρίες του Συμβουλίου και θέλουμε να συμμετάσχει και το τοπικό επίπεδο. με τη συμμετοχή των Ευρωπαϊκών Κέντρων Ενημέρωσης, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών. Άρα, πολλές πρωτοβουλίες θα διοργανωθούν σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα από όλους τους εταίρους μας. Το 2013, το έτος του πολίτη, θα αποτελέσει και προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Πολίτη. Και θα αποτελέσει προτεραιότητα και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα συνεργαστούμε στενά με την πρωτοβουλία Youth on the Move. Αυτό το λέω χάνει παραδείγματο. Άρα, το ανοιχτό και ευέλικτο αυτό πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους θα ενθαρρύνει πάρα πολλούς φορείς να συμμετάσχουν και να συμβάλλουν και αυτοί στο Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη. Κυρίε και κύριοι, προσβλέπω στη συζήτηση με εσά και στη συνεργασία άλλωστε μαζί σα για την πρωτοβουλία αυτή για το Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη για το 2013. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπίρνερτ. Πώ λέγεται, Μπερνέρτ, πώ λέγεται το όνομα Μπερνέρτ. Η συγκητής μας Χέφνερ θα θελήσει να παρέμβει μάλλον. Η αρμόδια από τη ουσίας επιτροπή είναι η ΛΥΜΠΕ που σκοπεύει να υιοθετήσει την έκθεσή της μέχρι τα τέλη Μαρτίου και περιμένει τη γνωμοδότησή μας στις 20 Μαρτίου. Μέχρι τις 20 Μαρτίου. Οπότε καλό θα είναι να συνεχίσουμε την εξέταση αυτού του θέματος 27 Φεβρουαρίου. Ας ακούσουμε τις πρώτες πατερίες του εισηγητού. Äh, Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε κυρία Περνέρ. Σήμερα θα θέλαμε εν συντομία να ενημερώσουμε τους συναδέλφους. Καταρχάς, ε, μας έκανε μια ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις προθέσεις της και μετά δική μου επιθυμία ως ε, μοναδικός υπεύθυνος και αρμόδιος για την Επιτροπή μας θα ήθελα να ακούσω και τα σχόλια των συναδέλφων, τις επιθυμίες ενδεχομένω των συναδέλφων και στην επόμενη συνεδρίαση θα σας παρουσιάσω ένα πρώτο σχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε το Μάρτιο. Και έτσι η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να μην λάβει ένα έτοιμο, προετοιμασμένο, τελειωμένο έγγραφο, αλλά εγκαίρως να μπορέσει να συμμετάσχει στην όλη διαδικασία. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα ε, να μην επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά γενικά να διαγράψω μία γραμμή, μία κατεύθυνση στην οποία θεωρώ ότι θα κινηθούν οι συζητήσεις οι οποίες έχουν γίνει ως τώρα προκειμένου το Ευρωπαϊκό Παϊκό Έτος για τον Πολίτη, το οποίο αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για μας και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ασφαλώς, αλλά και για την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ειδικά, να καταδείξουμε τη σημασία της Ενωμένης Ευρώπης για τον πολίτη. Και παράλληλα να καταστήσουμε σαφές αυτό που μας ανέφερε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρουσίαση του προγράμματος της, ότι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται και θα πρέπει να βρίσκεται ο πολίτης. Θα λάβει χώρα άλλωστε ένα χρόνο πριν από τις επόμενες ευρωεκλογέ. Και ελπίζω ότι σε αυτές τις εποχές όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση περνάει από σύνοδο σε σύνοδο και από μέτρα διάσωσης σε μέτρα διάσωσης, νομίζω ότι καλό θα είναι να αξιοποιήσουμε κατά το μέγιστο την ευκαιρία αυτή για να διευκρινίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε στον πολίτη ότι πραγματικά βρίσκεται στο επίκεντρο, στον πυρήνα της ε, πολιτικής ε, και όχι, δεν αποτελεί απλά έναν θεατή που κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα και παρακολουθεί αποφάσεις που λαμβάνονται ανταυτού. Άρα, πέρα από το, την πτυχή της ασφάλειας, ε, της, συγγνώμη, της ελευθερίας κίνησης και μετακίνησης, καλό είναι να δώσουμε μια επιπλέον διάσταση να δώσουμε τη διάσταση πιο έντονα της συμμετοχής στα διάφορα επίπεδα. Και σημαντικό είναι η επικοινωνία η οποία προγραμματίζεται να μην είναι μονομερής, να μην περιλαμβάνει μόνο ενημέρωση του πολίτη να μην περιλαμβάνει μόνο ευαισθητοποίηση του πολίτη. Όχι, να λάβουμε και αντίστροφα μέτρα. Μέτρα κατά τα οποία θα ρωτήσουμε τον πολίτη τι προβλήματα έχει, ποιε ιδέε έχει για το μέλλον τη Ευρώπη και θα κάτσουμε και θα ακούσουμε, θα εισακούσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη. Και ρόλο παίζει ασφαλώς το θέμα της νομικής βάσης. Θα πρέπει να κοιτάξουμε και τον προπολογισμό για την όλη διοργάνωση αλλά χαίρομαι σε κάθε περίπτωση. Θα χαιρόμουν να ακούσω και από τους άλλους συναδέλφους ε, τι στοιχεία θα τους ενδιαφέραν ιδιαίτερα για να προσθεθούν στην γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής μας. Όπως σας είπα την άλλη φορά, στην επόμενη συνεδρίαση θα σας υποβάλω και μια, ένα γραπτό σχέδιο. Ευχαριστώ κύριε Χέφνερ. Συνάδελφο Γκερέρο, Μπρόνς ζήτησαν το λόγο. Να ξεκινήσουμε με την κυρία τον κύριο Γκυρέρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. <coughs> Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά ταυτόχρονα ε, να πω ότι συμφωνώ και με όσα είπε και η Κομισιόν και ο κύριος Χέφνερ. Είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου αυτούς τους καιρούς που ζούμε, όπου πολλοί πολίτες απομακρύνονται από την Ένωση λόγω της οικονομικής κατάστασης, λόγω των δυσκολιών τις οποίες βιώνει η ολόκληρη Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε απευθείας στους πολίτες και να τους πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη είναι και ένα σχέδιο δικαιωμάτων, ηθαγένειας, ευκαιριών. Υπό την έννοια αυτή, η συνθήκη της Λισαβόνας έθεσε την ηθαγένεια στο επίκεντρο καταφέραμε να εγκρίνουμε την νομοθετική πρωτοβουλία για ε, την πρωτοβουλία των πολιτών και του χρόνου έχουμε και το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε ώστε στα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών που αυτή τη στιγμή διακατέχονται από άγχος και αγωνία να τους πούμε ότι η Ευρώπη παρέχει δικαιώματα, παρέχει και ευκαιρίες. Άρα, ο τρόπος με τον οποίο εστιάζει ο κύριος Χέφνερ, όπως πριν άλλωστε μας είπε και η Κομισιόν, είναι η κατάλληλη προσέγγιση. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην έμφαση που δίνει η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε την εστίασή μας, δηλαδή να αναφερθούμε στα δικαιώματα, τις ε, ευκαιρίες, την ενημέρωση από μια γενικότερη, ευρύτερη σκοπιά, που δεν θα μετατρέπει τους Ευρωπαίους πολίτες μόνο σε άτομα τα οποία μπορούν να μετακινούνται εντό της Ένωσης, αλλά εκεί που θέλουν να πάνε να βρουν και ευκαιρίες, να βρουν και δικαιώματα, τα οποία θα τους παρέχει η Ένωση. Στηρίζω λοιπόν και θα ρίνω τον κύριο Χέφνερ όταν θα εκπονεί στην γνωμοδότησή του προς την Επιτροπή Λίπε να είναι μια πιο πλήρης που να μην περιορίζεται μόνο στα θέματα της μετακίνησης, ελευθερίας μετακίνησης των πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Γκερέρο. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ πολύ. Οι πολίτες ορίζονται ως ε, μέλη ενός κράτους. Η έννοια πολίτης, αν θυμάμαι καλά, μπήκε ε, στη συνθήκη του Μάστριχ νομίζω και από το πρώτο σχέδιο είχε βγει η λέξη federal ε, μετά από τότε πρόταση του Πρωθυπουργού John Major που έλεγε ότι αν βάλουμε τη λέξη federal, ομοσπονδιακό, σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί ένα κράτο. Τέλο πάντων, τη λέξη πολίτη, ε, citizen, είτε δεν κατάφερε, δεν προσπάθησε να την ε, διαγράψει. Αλλά κατά την άποψή μου, όπως λέει και ο Τάμπιτ, ένας ε, Άγγλος πολιτικός, λίγο έτσι άκομψα, είπε ότι αν κάτι πλέει, κολυμπάει ως πάπια και κράζει ως πάπια, μάλλον είναι και πάπια. Άρα, αντίστοιχα, ο πολίτης, ο Ευρωπαίος, τι σημαίνει ότι ζει σε ένα κράτος ε, που έχει συγκροτηθεί, ένα κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση, αστικά. Έχουν, ε, πρέπει να πω, από τις περισσότερες ε, σημαντικές αποφάσεις ε, αποκλειστεί οι πολίτες. Παραδείγματο χάρη δεν έγιναν δημοψηφίσματα για τις συνθήκες που εγκρίθηκαν, αλλά τους δώσαμε ως αντάλλαγμα την πρωτοβουλία των πολιτών. Πρώτα απ' όλα, για να γίνει κάτι πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, κάτι αρκετά δύσκολο ή μάλλον πολύ δύσκολο για απλού πολίτε ή ε, μικρέ ομάδε πολιτών. Δεύτερον, αυτή η πρωτοβουλία μπορεί να απορριφθεί σε πολύ πρώιμο στάδιο, γιατί μπορεί να είναι κατά των ευρωπαϊκών αξιών, μπορεί να είναι επιφανειακή ή με απάντηση που πήρε τον κύριο Σεύκοβιτ, αν είναι και κατά των συμφερόντων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάλι μπορεί να απορριφθεί η πρωτοβουλία για αυτό το λόγο. Επομένω, η πρωτοβουλία των πολιτών δεν δίνει ουσιαστικά στους πολίτες πραγματική εξουσία, πραγματική δύναμη θα είχαν όμως πραγματική δύναμη αν ψήφιζαν μέσω των δημοψηφισμάτων πολίτε, αλλά αυτή τη δύναμη δεν τους τη δώσαμε. E Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Μπρόνση και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μίτα Μάκη. Όπως είπατε πράγματι οι πολίτες είναι στο επίκεντρο. Είναι το σημαντικότερο στοιχείο ο άξονα γύρω στον οποίο κινούνται τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Ένα θέμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η πρόσβαση στην ενημέρωση. Δεν θέλουμε να τους δώσουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να έχουν τη δυνατότητα να πούν τι θέλουν. Τώρα, τώρα που συζητάμε την πρωτοβουλία αυτή, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Έτσι δεν θα μιλάμε μόνο, δεν θα μένουμε στα λόγια, αλλά θα τους δώσουμε και πραγματική δύναμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδίως σήμερα. Γιατί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα έπρεπε. Και πρέπει κάτι να κάνουμε. Γιατί όταν έρθουν οι προσεχείς ευρωεκλογές και αν η προσέλευση είναι όπως ήταν και πριν, 30% θα έπρεπε αυτό να μας προβληματίσει, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Εμείς εδώ πώς μπορούμε να αποφασίζουμε εκ μέρους των ευρωπαϊκών πολιτών. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Πρόσβαση στην ενημέρωση. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία γιατί μόνο μετά από αυτό μπορούμε εμείς και οι πολίτες να πούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες προτάσεις και ούτω καθεξής. Grazie, se concludere questo dibattito il collega. ευχαριστώ. Κύριε Χέφνερ, θέλετε να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ε... ευχαριστώ. Συνάδελφε Κεραίρο για Μάκη Μπρόνς, άκουσα και σημείωσα τις, προ... τις προτάσεις που κάνετε για την πρόσβαση στα έγγραφα, για παράδειγμα. Θα καταθέσω μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση, να πω στον κύριο Μπρόντς ότι ναι, οι πολίτες βρίσκονται στον πυρένα της κοινή Ευρώπης, της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι πολλά πρέπει να κάνουμε ακόμα, προκειμένου αυτό να μεταφραστεί και να βιωθεί, αν θέλετε, στην πραγματικότητα αυτό το γεγονός. δεν ε, ωφελεί κανένα να είμαστε κοινικοί και αρνητικοί. Θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να ωφελήσουμε τον κόσμο καλύτερα. Και αν τα πάμε καλά, νομίζω ότι μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή με το Ευρωπαϊκό Έτος του Πολίτη. Θα ήθελα λοιπόν, αν οι άλλες ομάδες έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες θα ήθελα να δουν να αποτυπώνονται στο τελικό σχέδιο, να με ενημερώσουν μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, μάλιστα. Ευχαριστώ. 27 Φεβρουαρίου λοιπόν θα έχουμε στην ημερήσια διάταξη και πάλι το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών και ο συνάδελφος Χέφνερ θα μας παρουσιάσει μια ανέκτηση από τη βάση της οποίας θα είναι εύκολο να συνεχίσουμε την συζήτηση που σήμερα μόλις αρχίσαμε. Το σημείο 16 τώρα που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού, λαμβάνοντα υπόψη την εξέλιξη των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που αντιπροσωπεύουν τι εθνικέ κυβερνήσει μετά την έναρξη ισχύω τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Έκθεση Λαμασούρ. Ο συνάδελφο Λαμασούρ είναι παρόν. Θυμίζω ότι στι 22 Νοεμβρίου μα είχε παρουσιάσει ένα έγγραφο εργασία. Ζητήθηκε και μια ανέκθεση πρωτοβουλία, μάλιστα, πολύ έτσι ε, ευρέω σπάσματος και η έκθεση του κ. Λαμασούρα αφορά μια ε, ρύθμιση, μια τροποποίηση του κανονισμού σε σχέση με τις, σχέσεις, σε σχέση με τις επαφές με τα θεσμικά όργανα. Κύριε Λαμασούρ, μας ε, αναπτύξετε καλύτερα τη θέση σας εσείς ο ίδιος. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όντως, όπως το θυμήσατε κι εσείς, για το γενικότερο πρόβλημα των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και την ε, εκπροσώπηση των κυβερνήσεων, όπως προκύπτει από τη συνθήκη της Λισαβόνας και από την πρακτική που ακολουθείται εδώ και δύο χρόνια, Έχουμε εξ ονόματος τη ε, συνταγματική. έχετε μάλλον εσεί εξ τη Επιτροπή, ζητήσει από την διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να δεχτούν μια έκθεση πρωτοβουλία και μα ενημερώσαν ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, στην ε, συντακτική συνεδρίαση για το δεύτερο ήμιση της θητείας, η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θα ασχοληθεί με αυτό το αίτημα και πιθανότατα θα δώσει και θετική συνέχεια. Ε, εν τω μεταξύ, όπω είπατε, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα θέμα πολύ πιο περιορισμένο, που είναι όμως απαραίτητο. Ένα είδο χτενίσματο ε, του ιστορικού κανονισμού λειτουργία του Κοινοβουλίου, για να λάβουμε υπόψη τη συνθήκη της Λισαβόνα και το νέο ρόλο, ή εν πάση περιπτώσει της διευκρίνησης που γίνεται στη συνθήκη της Λισαβόνα για τον ρόλο του ε, Συμβουλίου σχέσεις δηλαδή ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και το συγκεκριμένο ζήτημα είναι η πίεση που μπορεί να... Οι ερωτήσει που μπορεί να θέσει οργανώνοντα συγκεκριμένε συνεδριάσει στην Κομισιόν και στο Συμβουλίο είναι μια παλαιότατη διαδικασία στην Ένωση και σήμερα ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι σε ένα μεγάλο τμήμα της ε, δραστηριότητάς του το Συμβούλιο βασικά είναι ένα νομοθετικό όργανο άνω βουλή ενός θεσμικού συστήματος με δύο βουλές και επειδή είναι διαφορετικό από το κοινοβούλιο αλλά σε ισότιμο επίπεδο Δεν χρειάζεται πλέον να τεθούν ε, ερωτήσεις ε, από το Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο. Θέλουμε να τροποποιήσουμε το άρθρο 116 παράγραφο 1, 2 και 5 έτσι ώστε να περιοριστεί η ώρα των ερωτήσεων σε ερωτήσεις που τίθεται προς την Επιτροπή, που είναι το εκτελεστικό σώμα εκτελεστική εξουσία και είναι απόλυτα θεμητό η νομοθετική εξουσία να μπορεί να θέτει όσες ερωτήσεις θέλει στην εκτελεστική. Ωστόσο προτείνεται να τροποποιηθεί επίσης το παράρτημα 2 του κανονισμού μας για να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι σε ορισμένους τομείς η εκτελεστική εξουσία ασκείται από τις εθνικές κυβερνήσεις και άρα από το Συμβούλιο. Οπότε πλέον δεν μπορούμε να θέσουμε ερωτήσεις στο πεδίο των νομοθετικών ζητημάτων, αλλά στο τομείς όπου διαπιστώνουμε ότι η εκτέλεση εξαρτάται από το Συμβούλιο και δεν είναι ικανοποιητική, τότε θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη δυνατότητα να θέτουμε ερωτήσεις. Πολύ συγκεκριμένο λοιπόν θέμα. Ένα είδος, όπως σας είπα, ε, καθάρεσης του δικού μας κανονισμού. Ο κύριος Γκερέρο ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ παρεμβαίνω στο όνομα της κυρίας Γκουρμάη που δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ παρούσα και είναι σκιώδης εισηγητής για αυτή την έκθεση. Εν γέννη θέλουμε, ε, θέλουμε να υποστηρίξουμε την θέση του κυρίου Λαμασούρ σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο το έχουμε ήδη συζητήσει και στους συντονιστές και σε άλλου είδους ε, συνεδριάσεις ότι ε, είναι αλήθεια ότι ε, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου θα πρέπει να γίνει μια πολύ ευρύτερη αναθεώρηση των σχέσεων ανάμεσα στο Συμβούλιο, στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο και ευρύτατο συζήτηση σε σχέση με το ρόλο του Κοινοβουλίου με δεδομένες της μεταρρύθμισης που γίνεται σε ορισμένες μορφές λήψη αποφάσεων στην της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτέλεσης αυτών. Ε, νομίζω λοιπόν ότι είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να κινηθούν παράλληλα δύο εκθέσεις, η αυτή του κυρίου Λαμασούρ και η άλλη για τον θεσμικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης. Γι' αυτό θα έχουμε την ευκαιρία στην Επιτροπή Αύκο να το συζητήσουμε ευρύτατα εγώ συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε ο κύριος Λαμασούρ. και τώρα για το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης που μας είπε ότι είναι ένα μικρότερο κομμάτι μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εν γέννη είμαστε υπέρ του να σταματήσουν αυτού του είδους ερωτήσεις που διατυπώναμε όταν η εξουσία του Κοινοβουλίου δεν ήταν αντίστοιχη με αυτήν του Συμβουλίου από άποψη θεσμική, ωστόσο να διατηρηθεί η δυνατότητα να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις όταν είναι ε, τα θέματα εκτός της νομοθετικής διαδικασίας όταν ε, υπάρχει πολιτικό ή στρατηγικό ενδιαφέρον και αξίζει το Κοινοβούλιο να συνεχίσει να, να, να, ασκεί τέτοιου είδους ελέγχο, μέσω των κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Υποστηρίζω εν γέννη λοιπόν τα όσα μας είπε ο κύριος Λαμασούρ και θυμίζω κάτι που δεν χρειάζεται καν να σας το θυμίσω γιατί είναι στο μυαλό όλων των μελών της Επιτροπής μας ότι δηλαδή αυτό αποτελεί μέρος ενός μικρού κομματιού μιας ενός ευρύτερου προβληματισμού που πρέπει να κάνουμε για τις σχέσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Ehm, Ο κύριος Νταφ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λαμασούρ για τις προτάσεις τις διατυπώνει και με τις οποίες φυσικά συμφωνώ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρέπει να πω επίσης ότι Περιμένω με πολύ μεγάλη ανυπομονησία να λάβω μέρος στις συζητήσεις ε, που θα έχουμε, τις πιο εκτεταμένες συζητήσεις, τις οποίες θα έχουμε όταν θα επανέλθει μετά τις κοινοβουλευτικές επαφές με τα Εθνικά Κοινοβούλια και το Συμβουλίο. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία 4. Στην ε, συγκεκριμένη αυτή τροπολογία αναφέρεστε σε ένα κριτήριο εδώ με αρνητικό τρόπο. Δηλαδή, τι εννοώ. Λέτε συγκεκριμένα ότι Δεν θα αμφισβητήσουμε το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές και δημοσιονομικές αρμοδιότητες. Κατά την άποψή μου θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια εναλλακτική προσέγγιση και να αναφερθούμε και σε κάποιες ε, αρμοδιότητες συντονισμού και πολιτική, άσκησης πολιτικής. Άρθρο 16.1. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να ορίσουμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο τις εκτελεστικές αρμοδιότητες του Συμβουλίου. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει το λιγότερο τουλάχιστον μια συζήτηση μεταξύ μου και του Συμβουλίου. Και θέμα αυτή τη συζήτηση θα ήταν ακριβώ. ο βαθμό ε, που η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, αλλάζει τι ε, εκτελεστικέ εξουσίε του Συμβουλίου. Αν ο κύριο Λαμασούρ έχει έντονα συναισθήματα επ' αυτού, πράγμα το οποίο είμαι σχεδόν βέβαιος, Παρ' όλα αυτά θα τον παρακαλέσω να την λάβει υπόψη και να την μελετήσει και αυτή την αναλλακτική προσέγγιση. Ρανζέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε Καζίνη. Θέλω να συγχαρώ τον Αλένα Λαμασούρ. the constitutional... Πιστεύω ότι στη συνταγματική προσέγγιση το Συμβούλιο έχει μια διτή φύση αν θέλετε. Δηλαδή, είναι ένα νομοθετικό σώμα και ως τέτοιο δεν θα πρέπει relations in all the countries that have two chambers. να θέτει ότι στο κοινοβούλιο Δεν χρειάζεται λοιπόν μια τέτοια διαδικασία, δεν είναι απαραίτητη. Αλλά δεν είναι αυτή η μόνη ιδιότητα του Συμβουλίου. Ιδίω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η διάσκεψη κορυφή των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Τέλο πάντων, το Συμβούλιο γενικά έχει και μια άλλη ιδιότητα, μια άλλη φύση, αν θέλετε, που θα την αποκαλούσα ένα θεσμό πολιτικής κατεύθυνσης, συντηρεί το πολίτικο που λένε και οι Ιταλοί. Συντηρεί το πολίτικο. Or uh, Ορίζει λοιπόν τους βασικούς στόχους της Ένωσης. Αυτή είναι η δεύτερη αρμοδιότητα του Συμβουλίου. Ένα ορισμό άκρο πολιτικό του έργου του Συμβουλίου είναι αυτό. Από αυτή την ιδιότητά του, αυτό το σώμα που έχει αυτό τον, το καθήκον του Ιντιρίτσο πολίτικο, αυτή τη πολιτική καθοδήγηση, πολιτική κατεύθυνση, εκεί μπορεί το κοινοβούλιο να έχει κάποιε σχέσει και να κάνει τι ερωτήσει του και να είναι να ζητά λογοδοσία ενδεχομένω. Έτσι μπορώ να το καταλάβω. Ίσως όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα ξανασκεφτούμε, να τα επανεξετάσουμε, να φτιάξουμε ένα καινούργιο θεσμικό πλαίσιο. Και θα μπορούσαμε να δούμε τότε αν το Συμβούλιο είναι ένα ομοσπονδιακό συμβούλιο πλέον, και τη θέση του Κοινοβουλίου. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. Συμφωνώ λοιπόν πλήρως με την προσέγγισή σας σε αυτό το θέμα. Αλλά βέβαια συμφωνώ και με την άποψη ότι θα μπορούσαμε πιθανότατα αυτές τις ιδέες να τις αναπτύξουμε για να προσπαθήσουμε να ορίσουμε με πιο συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο την προβλέψιμη εξέλιξη του θεσμικού μας πλαισίου. Και σε αυτή την περίπτωση δεν ενδεχομένως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ανάλυση που θα μας οδηγούσε ίσως σε ένα πιο ομοσπονδιακό, πιο ολοκληρωμένο όραμα. Σας συγχαίρω όμως γιατί η έκθεσή είναι πολύ ξεκάθαρη ως προς την διπλή αυτή φύση που θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά τη μία από την άλλη. Ευχαριστώ. Κύριε Λαμασούρ, μπορείτε να κλείσετε. Α, έχει άλλη παρέμβαση. Ο κύριος Χέφνερ. Äh, ναι, αλλά θα είμαι σύντομος. Γιατί φαίνεται ότι Ίσως να είναι μικρό το πρόβλημα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την μετέπειτα εξέλιξη της Ένωσης. Η δικτύωση των θεσμικών οργάνων και η προώθηση του θεσμικού διαλόγου από πλευρά μας. Υποστηρίζουμε τις ε, απόψεις του κ. Λαμασούρ. Από πολιτικής άποψης δεν βλέπουμε να υπάρχει ανάγκη αλλαγή τη πορεία. Θεωρούμε ότι σωστά έχει γίνει η επεξεργασία του προβλήματο και σωστέ είναι και οι προτάσει που έχουν κατατεθεί. Μάλιστα. Κύριε Λαμασούρ, θέλετε να ολοκληρώσετε αυτή τη συζήτηση. President. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Ο Παόλο Φανζέλ έλεγε δικαίω ότι έτσι όπως έχουν ε, τα πράγματα. Ε, ο συνάδελφό μα ο Ντάκ πριν από, ο Μπρόνς πριν από λίγο χρησιμοποίησε την παρομοίηση με την πάπια. Εντάξει, μια πάπια είναι μια πάπια, αλλά το Συμβούλιο είναι ένα κάστορα. Ξέρετε ότι το Μεσαίωνα θεωρούσαν ότι μπορούσε κανείς να τρώει την Παρασκευή κάστορα, γιατί επειδή ζούσε στο νερό, θεωρεί το ψάρι από γαστρονομικής άποψης. Ταυτόχρονα όμως είναι θηλαστικό κτλ. Αλλά, εν περιπτώσει, το... ε, πάλι καλά που δεν τρώγανε και νυχτερίδες. Ε, το Συμβούλιο είναι κάστορας, λοιπόν. Αν λοιπόν ε, το Συμβούλιο είναι ψάρι και εμείς έχουμε το δικαίωμα να, να διαλεγόμαστε μαζί του υποβρυχίως και όχι χερσαίος. Ε, πολύ δυναμικά, όμως πρέπει να το εκφράσουμε αυτό και με αρνητικό τρόπο όπως το προτείνω στο κείμενό μου παραμένοντας όμως πολύ αυστηρή από νομικής άποψης ε, να το μπορούμε να το εκφράσουμε και θετικά, με θετικό τρόπο, στο λέει και ο Άντρογο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μπορούμε να δούμε με τους συναδέλφους να δώσουμε κάποιο πιο θετικό τόνο στην τροπολογία 4 με την προϋπόθεση όμως υπό τον όρο ότι το κείμενο θα είναι νομικώς ακριβές και η μεγάλη συζήτηση την οποία ονειρεύεται ο Άντριου και εγώ ίδιος και πολλοί από εμά για την πραγματική φύση αυτού του μυστήριου ζώου και εν γέννη πώς καλύτερα θα οργανώσουμε επί τη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας και μέσα στο σημερινό πλαίσιο τις σχέσεις μας με αυτό το άλλο θεσμικό όργανο, πρέπει λοιπόν την ουσία, τη συζήτηση ουσίας να την παραπέμψουμε σε μια έκθεση πρωτοβουλία τις οποίες υποστηρίζουμε την εκπόνηση. Ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ. Άρα λοιπόν, τι μένει, προθεσμία για υποβολή τροπολογιών και μέρα για την ψηφοφορία. Πρόταση της Προεδρίας είναι τροπολογίες να μπορούν να υποβληθούν μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου το μεσημέρι και η ψηφοφορία να γίνει στις 28 Φεβρουαρίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις, μπορεί να γίνει αυτό και να περάσουμε και στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης που αφορά την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολίτων. Η κυρία Γκουρμάη δεν μπόρεσε να βρίσκεται στις Βρυξέλλες, να φτάσει στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι ακόμα και χτες βρισκόταν ε, στην Κωνσταντίνα. Αλλά έχουμε τον συνάδελφο Λαμασούρ εδώ που μπορεί να μας ε, ενημερώσει για αυτή την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για αυτό το θέμα.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 Α, δεν μπορούσε να είναι παρούσα γιατί είχε ανελημμένες υποχρεώσεις. Δεν θα έρθει εκείνη, αλλά υπάρχουν στην αίθουσα ή θα έρθουν στην αίθουσα μέλη της Επιτροπής Αναφορών τόσο από τους σοσιαλιστές όσο και από τους πρασίνους αλλά και από το ΕΛΚΑ. Ο κύριος Μποστινάρου, ο κύριος Μποστινάρο από τους σοσιαλιστές, η Όκεν από τους πρασίνους και η Τσέβα από το ΕΛΚΑ περιμένουμε, φτάνουν. Bene, allora io pregherei il collega Lamassur Μάλιστα. Λοιπόν, να παρακαλέσω τον κύριο Λαμασούρ να μας παρουσιάσει την κατάσταση. Κύριε Πρόεδρε, εγώ στα ζηταγά σας, αλλά για αυτή την έκθεση δεν είμαι συνεισηγητής. Οι σχέσεις μου. Ε, κάθε είδους σχέση είναι πολύ ανεπτυγμένη με τη Ζήτα Γκουρμάη, αλλά δεν τα κάνουμε και όλα χέρι-χέρι. Ε, εγώ είμαι σκιώδης της ομάδας μου, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στην ΑΦΚΟ, αλλά ε, από ό,τι ήθιστε, αν λείπει η ε, ένα μέλος της ομάδας του συνήθως είναι ο εκπρόσωπός του. Εγώ φυσικά να δώσω τη γνώμη μου, αλλά δεν θέλω να ξεπεράσω τα δικαιώματά μου. Bueno. Eh, Θέλω να αποφελθώ της τελευταίας, όχι αυτή, αλλά της τελευταίας στην προηγούμενη συζήτηση παρά του κ. Αμασούρ, για να πω ότι πιστεύω ότι αυτή η συνεδρίαση σε επιτροπή θα είναι η τελευταία στην οποία θα είμαι συντονιστής της σοσιαλιστικής ε, ομάδας. θα καταλήψω την αρμοδιότητα αυτή, διότι εξελέγει αντιπρόεδρος στην ομάδα μου. Δεν το λέω για να σας το αναγγείλω αυτό απλά, απλά για να σας επισημάνω ότι όπως ε, έχετε ίσως διαπιστώσει τους τελευταίους μήνες και εγώ κάστορα είμαι. Άλλοτε είμαι ψάρι, άλλοτε είμαι κρέας, άλλοτε είμαι λαχανικό, άλλοτε είμαι φρούτο, <laughs> διότι περνάω από το ένα θέμα στο άλλο καθότι τα μέλη της Επιτροπής μου μου ζητούν να τους αντικαταστήσω για τις διάφορες εκθέσεις. Είμαι λοιπόν και χορτοφαγικός και ο προκυπευτικός κάστορας. Το συγκεκριμένο όμως ε, σημείο, όποια και αν είναι η τόσο αναπτυγμένη σχέση μεταξύ του κ. Λαμασό και της κυρίας ε, Γκουρμάη, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι υπάρχει μια κοινή θέση στην Επιτροπή αυτή. Δηλαδή ότι εργαζόμαστε από κοινού με την Επιτροπή Αναφορών, αλλά δεν θα τους δώσουμε και την, τα πρωτεία, την ηγετική θέση ό,τι αφορά την ακρόαση ή την, ε, τον καθορισμό των διαδικασιών για την ε, πρωτοβουλία των πολιτών, υποδοχή των αναφερόντων στο Κοινοβούλιο κτλ. Κάθε σεβασμό τρέφω βέβαια στην Επιτροπή Αναφορών και έχω και την καλύτερη δυνατή διάθεση να βρούμε τρόπους να εργαστούμε από κοινού στο θέμα αυτό, αλλά πάντα πρέπει να πω ότι θα προασπίζουμε τη θέση της ΑΦΚΟ ως Ηγέτηδο ή συνηγέτηδο επιτροπή τουλάχιστον, σε ό,τι αφορά τα θέματα που άπτονται τη πρωτοβουλία των πολιτών. Κύριε Λαμασούρ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ο συνάδελφος Γκερέρο, αυτή η συνηγετηδο επιτροπη τουλαχιστον σε οτι αφορα τα θεματα που απτονται της πρωτοβουλια των πολιτων κυριε λαμασουρ ευχαριστω κυριε προεδρε οπως ο συναδελφος γκερερο αυτη η επόμενη προσαρμογή του εσωτερικού κανονισμού έχει ως στόχο να ορίσει ε, τις προποθέσεις από τις οποίες το Κοινοβούλιο θα οργανώσει την δημόσια ακρόαση των ε, υπεύθυνων πρωτοβουλίας πολιτών που κατάφεραν να δρομολογήσουν τη σχετική διαδικασία. Θα θυμάστε ότι η Επιτροπή μας εργάστηκε σκληρά. Το τελικό κείμενο του κανονισμού για την πρωτοβουλία των πολιτών πολλά οφείλει στις ε, τροπολογίες της Επιτροπής μας. Αυτό το οποίο θελήσαμε ήταν κάθε πρωτοβουλία των πολιτών που έχει έρθει σε αισιοπέραση, έχει πετύχει δηλαδή. Δηλαδή, έχει συντάξει ένα κείμενο που είναι και συμβατό με τις αρχές της Ένωσης που φέρει την υπογραφή τουλάχιστον ενός εκατομμύριου πολιτών, τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών. Πριν η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, αποφανθεί για τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί σε αυτή την πρωτοβουλία, αποφασίσαμε να γίνει η δημόσια ακρόαση, την οποία θα οργανώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα λοιπόν που τίθεται σήμερα είναι πώς θα γίνει αυτό στην πράξη. Η τα Γκουρμά και εγώ το σκεφτήκαμε μετά από την κοινή έκθεση που είχαμε συντάξει για το σχέδιο κανονισμού. Η κυρία Γκουρμάη είχε επιφορτιστεί με την εκπόνηση μιας μικρής έκθεσης και συμφωνώ μαζί της απόλυτα. Φαντάζομαι ότι και η ομάδα μπορεί να το στηρίξει αυτό που θα πω ότι η διαδικασία, η πολύ απλή που προτείνεται, είναι αποδεκτή. Η ιδέα είναι να διατηρηθεί το πνεύμα της απλότητας που διαπνέει και όλες μας τις τροπολογίες στο σχέδιο κανονισμού. Για να τα πω πιο απλά και για να είναι πιο απλά τα πράγματα, κάθε φορά που θα έχει έρθει θέση ο πέρας, ε, θα έχει ευοδοθεί μια πρωτοβουλία των πολιτών και θα έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Μητρό που θα έχει ανοίξει την πρωτοβουλία αυτή, τότε την προκειμένη στιγμή εγγράφεται στη μερίσια διάταξη ή εν λόγω πρωτοβουλία στη διάσκεψη των πρόεδρων των επιτροπών. Ανάλογα με το θέμα, η διάσκεψη των πρόεδρων των επιτροπών αποφασίζει ποια θα είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπενθυμίζω ότι η πρωτοβουλία των πολιτών πρέπει να αφορά ένα νομοθετικό θέμα και επομένως 9 στις 10 τουλάχιστον η επιτροπή που θα επιλέγει η διάσκεψη των πέντε των επιτροπών θα είναι μία από τις νομοθετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου μας. Τώρα, επιτροπή που θα έχει την αρμοδιότητα για την διοργάνωση της ακρόασης θα πρέπει να έρχεται φυσικά σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενδεχομένως και με, άλλες, ε, με άλλους ε, οργανισμούς και θεσμικό όργανα για να οργανωθεί η δημόσια αυτή ακρόαση στην πράξη. Γιατί με τους άλλου οργανισμούς και θεσμικά όργανα. Γιατί με βάση τα θέματα η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, ίσως και άλλοι οργανισμοί, θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται ή να αφορώνται, αν θέλετε, από το θέμα αυτό, οπότε θα μπορούσαν να προσκληθούν και να θέσουν τα ερωτήματά τους και τις απόψεις τους. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα. Προβλέπεται μια τρίμηνη προθεσμία. Και όπως είπα η αρμόδια επιτροπή είναι αυτή η οποία θα προσκαλέσει είτε τους οργανωτές τη πρωτοβουλία των πολιτών, είτε μια αντιπροσωπεία τους, να έλθουν να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους στο πλαίσιο μια δημόσιας ακρόασης. Αυτή είναι η βασική αλλαγή και προσθήκη στον κανονισμό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη εδώ και μια άλλη ανησυχία. Μια άλλη μέρη. Ε, το συζητήσαμε μάλιστα διαμακρών κατά την εκπόνηση του κανονισμού αυτό το θέμα. Τι κάνουμε λοιπόν με πρωτοβουλίες που δεν πέτυχαν, δεν ευωδόθηκαν μεν, αλλά από πολιτικής πλευράς εκπροσωπούν, αντιστοιχούν σε ένα διάβημα το οποίο απαιτεί κάποιο είδους απάντηση, αντίδραση. Παραδείγματο χάρη, μια πρωτοβουλία που μπορεί να σκέντρωσε 900.000 υπογραφές, που να έχει να κάνει με ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο για την κοινή γνώμη, αλλά δεν έφτασε στο 1 εκατομμύριο υπογραφές. Ή να έχουμε 4 εκατομμύρια επιγραφές για μια πρωτοβουλία, αλλά να μην ε, συμπληρούνται ο ρυθμός των κρατών μελών, να λείπει ένα κράτος μέλος. Θα κυριαρχήσει ο νόμος της ιοποίησης, σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκολο. Έπρεπε να βρούμε μία απάντηση. Ε, μία φόρμουλα που μας φάνηκε ενδιαφέρουσα είναι να λαμβάνεται υπόψη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά με βάση της πολύ γνωστής και καλά δοκιμασμένης διαδικασίας του Κοινοβούλιο που είναι η διαδικασία των αναφορών. Άρα τότε θα είναι η Επιτροπή Αναφορών αυτή η οποία, αν το κρίνει σκόπιμο και χρήσιμο βέβαια, θα καλείται να δώσει μια συνέχεια σε αυτές τις πρωτοβουλίες που δεν κατέληξαν και θα αποφασίζει η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή των Αναφορών, ε, σύμφωνα και με τον ιστορικό κανονισμό του Κοινοβουλίου, τι συνέχεια θα δώσει και ποιε διαδικασίε θα ακολουθήσει. Αυτά ήταν γρήγορα γρήγορα τα στοιχεία που προτείνουμε στον κανονισμό προσθήκη ή τροποποίηση για να ε, ικανοποιήσουμε και τους ε, οργανωτές των πρωτοβουλίων των πολιτών και για να λάβουμε υπόψη και το σημαντικότερο δηλαδή τις σα πρωτοβουλίες αλλά και τι πρωτοβουλίε που δεν κατάφεραν να ο πέρας αλλά για τι οποίε χρειάζεται ένα είδο πολιτική αντίδραση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας που ήταν τόσο ε, ακριβείς όπως συνήθως και τώρα θα δώσω το λόγο σε κάποιον από τους εκπροσώπους της, μάλλον στους εκπροσώπους της Επιτροπής ε, Αναφορών. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπουλό. Να... Καταρχήν συμφωνώ με τα όσα είπε ο συνάδελφος Λαμασούρ, ωστόσο θα ήθελα εδώ να σας αναφέρω σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν και το αίσθημά μας ε, στην Επιτροπή των Αναφορών. Εμείς ε, δεν ζητήσαμε την, ε, να έχουμε την αποκλειστικότητα και την ε, προτεραιότητα. Αναγνωρίζουμε την ε, προτεραιότητα της ΑΦΚΟ, είναι προφανές αυτό, ωστόσο δεν θέλουμε να είμαστε εκτός από τις διαδικασίες της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών. Στο βαθμό που έχουμε σχετική εμπειρία θα θέλαμε λοιπόν να συνδεθούμε με τις δημόσιες ε, κροάσεις για αυτές τις ε, ε, πρωτοβουλίες που έχουν συγκεντρώσει ένα εκατομμύριο υπογραφές στα 3, στο 1 τέταρτο των κρατών μελών και ότι έχουμε τη συνήθεια να ασχολούμαστε με τέτοιου είδου αναφορές. Βεβαίω είναι πολύ ευρύτερε σε μέγεθο από αυτέ που συνήθω μα απασχολούν στην Επιτροπή Αναφορών, ωστόσο όσον αφορά την μορφή ακούγοντας τον Αλένα Μασούρ που λέει ότι αυτές που έχουν ε, ε, ας πούμε ένα εκατομμύριο υπογραφές αλλά ένα κράτος λιγότερο ότι θα πρέπει να εξετάζονται από την Επιτροπή Αναφοράς επειδή της είναι δύσκολο να προληφθεί κάτι τέτοιο στο βαθμό που γιατί η Επιτροπή Αναφορών να είναι ξαφνικά αρμόδια για να εξετάσει μια αναφορά 299.999 πολιτών ή όπου, όπου, τέσσερα, όπου το 1 τέταρτο των κρατών μελών έχει συνυπογράψει, συμμετέχει μάλλον, γιατί να είμαστε αρμόδιοι για αυτή την αναφορές ενώ όχι για τις άλλες. Για μας δεν είναι λοιπόν λογικό να μην ε, συμμετέχουμε εξ αρχής στις ακροάσεις της πρωτοβουλίας των πολιτών και επιθυμούμε όχι να έχουμε την αποκλειστικότητα, το επαναλαμβάνω, αλλά να συμμετέχουμε εξ αρχή σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι ώστε η Επιτροπή σα, σε συνεργασία με τη δική μα, να κάνει αυτό το αίτημα προ την διάσκεψη των Προέδρων που θα πρέπει να αποφασίσει για την απονομή των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας επιτροπής ε, για το θέμα. Υπάρχουν παρόντα και άλλα μέλη της Επιτροπής Αναφορών και πιστεύω πως θα ήταν ε, ενδιαφέρον να έχετε, ακούσουμε την άποψή τους για αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω πως ε, αυτό είναι μια πραγματική επιθυμία να είμαστε κι εμείς μετέχονται σε αυτή τη διαδικασία της πρωτοβουλίας των πολιτών. Αν είναι απογοήτευση, αν απογοητευτείτε από την Επιτροπή Αναφορών, να το ξανασυζητήσουμε. Αλλά εφόσον και εμείς ε, έχουμε αναφορές ε, που ασχολούνται με θέματα που θα μπορούσαν να καταλήξουν σε νομοθετικά κείμενα που δεν έχουν την απαραίτητη ευρύτητα, εύρος μάλλον. Ε, και έτσι θα μπορέσουμε όταν θα ασχοληθούμε με αυτές τις μικρότερες ε, εντός εισαγωγικών αναφορές να μπορέσουμε να δώσουμε μια επιπλέον απάντηση, απάντηση εφόσον θα έχουμε συμμετέχει στην ακρόαση μιας πρωτοβουλίας των πολιτών. Μια αναφορά στις πρωτοβουλίες των πολιτών. Νομίζω πως κάτι τέτοιο θα ήταν λογικό. και κυρίως θα στήριζε και την Επιτροπή Αναφορών, της Εργασίας της Επιτροπής Αναφορών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο τώρα η κυρία Όκεν. Άουκεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δώσατε και χρόνο για να μιλήσουμε. Θα εργαστώ εγώ για το θέμα αυτό και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν συμφέρει την Επιτροπή Αναφορών να καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις. Φυσικά θα τα βγάλουμε πέρα, όπως και να έχει. Δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ και για τον οποίο υποβάλλουμε αυτή την τροπολογία. Πιστεύουμε ότι αυτή η πολύ σημαντική ε, πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει να ακολουθήσει μια βασική διαδικασία στο Κοινοβούλιο. Είμαστε συνηθισμένοι στην Επιτροπή Αναφορά να συνεργαζόμαστε με τους πολίτες, αλλά ασφαλώς θα πρέπει να διαχωριστεί από το συνηθισμένο μας έργο, από τις αναφορές. Θα πρέπει να είναι η πρωτοβουλία των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σταθερή βάση, μια σταθερή επιτροπή στην Επιτροπή που θα έχει εμπειρία πάντα σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή ασφαλώς αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια δίκαιη και ίση αντιμετώπιση και γι' αυτό λοιπόν και υποβάλαμε αυτή την τροπολογία στην εξαιρετική σας έκθεση για να δοθεί πιο πολύ μεγάλη διαφάνεια και να υπάρχει ασφάλεια στην όλη διαδικασία και θα θέλαμε αυτό να μπει στην ατζέντα του Κοινοβουλίου και στη δική μας ατζέντα τρεις-τέσσερις μέρες πριν από κάθε φορά και πριν από την ακρόαση για να είμαστε βέβαιοι ότι σε κάθε περίπτωση θα έχουμε το χρόνο να, να επεξεργαστούμε το θέμα, να κυρώσουμε ενδεχομένω και τι ακροάσει εφόσον δεν είναι απαραίτητες. Άρα σας καλώ να μην το κάνετε αυτό προς όφελος της Επιτροπής Αναφορών, αλλά προς όφελος όλη τη πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών. Κάνουμε άλλο τόσο πολλά για να πείσουμε τους πολίτες μας για το τεράστιο βήμα προς τα εμπρός που σήμαινε η συνθήκη της Λισαβόνας και η πρωτοβουλία αυτή. Και πραγματικά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που εργάζεται με εξαίρετο τρόπο. Χρωστάμε στον πολίτη να υπάρχει μια σταθερή διαρκής δομή η οποία πάντα θα αναλαμβάνει την ευθύνη ασφαλώς βέβαια με συνεργάτη την εκάστοτε αρμόδια επιτροπή. Αυτό κρύβεται πίσω από την τροπολογία. Ελπίζω να σας βρει σύμφωνους η τροπολογία αυτή. Δεν βλέπω να υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων. Το θέμα είναι απλά να υπάρχει συμπληρωματικότητα στην εργασία μας. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Χέφνερ. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα... Να ευχαριστήσω όσους και να συγχαρώ όσους συνεργάστηκαν για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Πολιτών. Θα ήθελα όμως ε, σήμερα κατ' εξαίρεση να ξεκινήσω με ένα παράπονο γιατί αυτή η καλή συνεργασία που ε, χαρακτήρισε την αρχική φάση δεν συνεχίστηκε. Υπήρχε μια ομάδα τεσσάρων ατόμων από δύο επιτροπές, ε, από τέσσερις ομάδες, οι οποίοι κατήρθησαν την έκθεση αυτή από κοινού και θα συμφωνήσει άλλωστε και ο συνάδελφος Λαμασούρ, δεν είναι εδώ η κυρία Γουόλης και η κυρία Γκουρμάη δυστυχώς. δεν κάναμε τίποτα επέσχυδο, τίποτα ε, επέσχυδες ε, διαπραγματεύσεις. Όχι. Με πολύ υπομονή συζητήσαμε μεταξύ μας και για κάθε περίπτωση καταλήξαμε στην καλύτερη λύση. Επιθυμία μου θα ήταν να συνεχιστεί αυτό. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό εδώ. Ακόμα και μετά από την έκκληση των επικεφαλής της ΑΦΚΟ Okay, danke. Es es kann immer nur einer <laughs> reden. Äh, also es war dieses Gespräch allen Bitten zum Trotz nicht mehr möglich. Und jetzt haben wir eine merkwürdige. Και βλέπουμε λοιπόν μια περίεργη κατάσταση να διαμορφώνεται πλέον. να συμμετέχουν διάφορες ομάδες οι οποίες έχουν και εκπροσωπούν διάφορα και διαφορετικά συμφέροντα. Απευθύνω μια έκκληση να βρούμε κοινό τόπο. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα δυνατό αυτό και μάλιστα ε, είναι προς όφελος της πρωτοβουλίας των Ευρωπαίων πολιτών σε ό,τι αφορά την διοργάνωση των ακράσεων. Πρόκειται κάτι το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της πρωτοβουλίας των πολιτών. Επί ένα έτος συλλέγουν ένα εκατομμύριο υπογραφές οι πολίτες για να πετύχουν τελικά τι, μία ακρόαση, να εισακουστούν συμφωνήσαμε ότι η ακρόαση αυτή θα πρέπει να είναι μια ακρόαση στην οποία θα συμμετέχουν και το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εισακούσουν τις προτάσεις των ε, πολιτών. Όλα τα υπόλοιπα όμως έχουν μείνει ανοιχτά. Ποιος θα το διοργανώσει για παράδειγμα. Ποιες, ε, ποιοι όροι θα πρέπει να πληρούνται. Όλα αυτά ρε, δεν ρυθμίζονται στον κανονισμό. Με την ρύθμιση και την αλλαγή του κανονισμού από πλευράς του κυρίου Λαμασούρ και της κυρίας Γκουρμάη απαντώνται κάποια ερωτήματα, όχι όμως όλα δυστυχώς. Και αυτή η πρόταση μου προκαλεί και καινούργιες ερωτήσεις και καινούργιες ανησυχίες. Συγκεκριμένα, στην πρόταση αυτή η ιδέα είναι το, η πρωτοβουλία να απευθυνθεί στον πρόεδρο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών και μετά ο πρόεδρος της διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών να αποφασίσει ποια είναι η αρμόδια επιτροπή. Στη συνέχεια, ελέγχει η αρμόδια επιτροπή κατά πόσον πληρούνται όλοι οι όροι που θα πρέπει να πληρούνται από την πρωτοβουλία των πολιτών. Δηλαδή, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, η Επιτροπή Σταματικών Υποθέσεων, ανάλογα. Κάθε Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει και να αναπτύξει αυτή την αρμοδιότητα του ελέγχου. Και αυτό οι Επιτροπές θα το πετύχουν σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με την εμπειρία που έχουν, ανάλογα με το δυναμικό που έχουν οι γραμματείες τους. Εγώ θα ήθελα το Κοινοβούλιο να έχει μια διαρκή, ένα διαρκέ σημείο επικοινωνίας, να υπάρχει κόσμος ο οποίος να ξέρει τι θα πρέπει να ελέγχεται κάθε φορά και πώς θα πρέπει να διοργανώνεται η ακρόαση κάθε φορά. Δεν είναι μία κανονική συνήθις εκδήλωση του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός με, με τα άτομα που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία για να ξέρουμε Πόσοι θα έρθουν, ποιοι θα έρθουν, τι έξοδο ταξιδίου θα πρέπει να υπολογίζουμε. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός μορφοτύπος. Δεν είναι μια συνηθισμένη συνεδρίαση επιτροπής και θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα άτομο το οποίο θα έχει εμπειρία με αυτά τα πράγματα. Στο Γερμανικό Κοινοβούλιο με αυτούς που συνομίλησα μου είπαν ότι αν ε, υπάρχει κάθε φορά μια διαφορετική γραμματεία, μια διαφορετική επιτροπή, διαφορετικά άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα και την διοργάνωση θα έχουμε προβλήματα. Είπε η Επιτροπή Αναφορών τώρα να την διοργανώσουμε εμείς. Συμφωνώ ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι η Επιτροπή που έχει την εμπειρία στη συναστροφή με τους πολίτες, αλλά οι ειδικέ αρμοδιότητες θα χρησιμοποιούσαν οι ειδικέ ικανότητες των ειδικών επιτροπών. Και δεν θα ήθελα η συζήτηση να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να υποστηρίζει τη δική του επιτροπή. Καταλαβαίνω το πνεύμα των προτάσεων και θεωρώ ότι μία λύση θα ήταν να υπάρχει μία ενιαία ε, υπηρεσία στο Κοινοβούλιο. Θα μπορούσε να είναι η γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών. Και κατά τα άλλα, οι ακροάσεις να διοργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν και να απαντούν και να καλούν στις εκφράσεις αυτές η Επιτροπή Αναφορών και η αρμόδια Επιτροπή εκάστοτε μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά θα ήθελα να τα πω αυτά ανοιχτά στην Επιτροπή μετά από συζήτηση με τους εμπλεκόμενους και τους ενδιαφερόμενους. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν θα ήταν δυνατόν οι εισηγητές ε, οι οποίοι κατήρτισαν μια τόσο τέτοια θαυμάσια έκθεση να κάτσουν μαζί με την Επιτροπή Αναφορών και να προσπαθήσουν να βρουν μια κοινή λύση. Θα και θα θεωρούσα ότι θα ήταν αξιοθαύμαστο το έτος που θα ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία των Προελτών να υπερψηφίσει το Κοινοβούλιο τις σχετικές ρυθμίσεις με την ίδια συντριπτική πλειοψηφία που είχε υπερψηφίσει την ε, πρωτοβουλία και όχι με μια οριακή πλειοψηφία. Αυτή θα ήταν η δική μου έκκληση. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Γουερέρο, γιατί μετά πρέπει να φύγει και ζήτησε να παρέμβει λίγο νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Επειδή πράγματι πρέπει να φύγω, ήθελα να απαντήσω στα όσα άκουσα. Εγώ γενικά συμφωνώ με την ιδέα. Με πολλές γενικές ιδέες συμφωνώ. Δηλαδή, ότι πρέπει Το Κοινοβούλιο πρέπει να εργαστεί ως ένα όλο, ένα σύνολο και να μην ε, επιδιώκει κατακαιρματισμό σε διάφορε επιτροπέ, ιδίω για αυτό το θέμα τη πρωτοβουλία των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, εμεί είμαστε η επιτροπή που έχουμε μεν ε, εμπειρία, αλλά αυτοί που έχουν εμπειρία πιο πολύ συγκεκριμένη πάνω στο θέμα τη κοινότητα με είναι η Επιτροπή Αναφόρων και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Συμφωνώ και με αυτό που είπε ο κύριος Χέφνερ, ότι η συγγήτρα, ο οι Καλό θα ήταν να συνεδριάζουν μαζί με την Επιτροπή Αναφορών για να δουν ποιοι κοινοί χώροι, αν θέλετε, δράσεις υπάρχουν. Να ενημερωθεί η κυρία Γκουρμάη για το πώς ε, εξελίχθηκε αυτή η συζήτηση, να της μεταφέρουμε τα επιχείρηματα που ακούσαμε και πριν οριστικοποιήσουμε την άποψή μας, να έχουμε με επαφή με την ε, Επιτροπή Αναφορών, για να προσπαθήσουμε από κοινού να καταλήξουμε σε μια θέση η οποία θα αξιοποιεί, θα εκμεταλλεύεται την εμπειρία της Επιτροπής Αναφορών σε ό,τι αφορά την οργάνωση τέτοιων ακροάσεων, αλλά που επίσης, σύμφωνα και με αυτά που είπε ο κ. Λαμασούρ, να διατηρηθεί η ουσία της έκθεσης όπως αυτή τη στιγμή έχει συνταχθεί. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη γιατί θα πρέπει να πάω και σε μια άλλη συνεδρίαση. Αλλά καταρχά, ναι, υποστηρίζω την πρόταση. Είναι πολύ καλή και νομίζω ότι είναι σημαντικό να εμπλέκονται και τα Εθνικά Κοινοβούλια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα ζητήματα αυτά. καταλαβαίνω ότι θα προκύψουν ε, ενδεχομένω δυσκολίε κατά το μέλλον. Η πρωτοβουλία των ε, πολιτών είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά επί του παρόντος δεν γνωρίζω να υπάρχει καμία χώρα που να έχει να παρουσιάσει μια έτοιμη συνταγή. Η Ελβετία βέβαια ακολουθεί διαφορετικό σύστημα, αλλά γενικά σε όλες τις χώρες ε, είχαν, ε, όποτε είχαν τεθεί τέτοιες πρωτοβουλίες, είχαν απορριφθεί από τα κοινοβουλία. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει Αν αποτύχουν οι πρώτες 5-6 τέτοιες πρωτοβουλίες, δεν θα έχει νόημα να συνεχιστεί η πρωτοβουλία, γιατί θα θεωρήσει ο πολίτης ότι δεν εισακούεται. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε με ποια αιτιολογία θα γίνει η μη αποδεκτή μια τέτοια πρωτοβουλία. Γιατί εδώ έχουμε μια πραγματικά απίστευτη ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω λοιπόν εδώ να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας εδώ. Αν δεν προετοιμαστούμε καλά, τελικά θα καταλήξει, αν θέλετε, στον κάβο των αχρήστων αυτή η πρωτοβουλία. Θα ξεχαστεί. Λυπάμαι που εξέφρασα τόση πολύ απεσιοδοξία, αλλά νομίζω ότι καλό είναι όλα αυτά να τα σκεφτούμε εκ των προτέρων και όχι των υστέρων. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι σύντομη, δεν θέλω να επαναλάβω ε, συμφωνώ με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι τη Επιτροπή Αναφορών. Θέλω να επιστήσω την προσοχή σε τρία πράγματα. Καταρχήν να θυμίσω ότι ε, καταρχήν ε, η οι συγητέ και οι σκιώδες συγητής έχουν συνεργαστεί για αυτή την ε, πρωτοβουλία και εδώ κάνω έκκληση ώστε η καλή ε, συνεργασία που είχαμε τους τελευταίους μήνες να διατηρηθεί ε, και αυτό με όλο το σεβασμό στις, και στις δυο μας επιτροπές. Και όσον αφορά τις αναφορές που πέτυχαν ή που απέτυχαν από την άποψη την τυπική, εμείς ποιο μήνυμα στέλνουμε ανάμεσα σε δύο ομάδες επιτροπών, δηλαδή τις επιτροπές που ασχολούνται με τα επιτυχημένα και αυτές που, με το, που ασχολούνται με τα αποτυχημένα. Είναι ένα μήνυμα και προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, ξύριμα θα ξέρουν και εκείνοι θα καταλάβουν πώς ε, πρέπει να ενεργήσουν για να έχουν μια πετυχημένη πρωτοβουλία. Θα πρέπει να κρατήσουμε αυτό το πράγμα ότι όλες οι επιτροπές έχουν τη σημασία τους και θα πρέπει να έχουμε ένα ενοποιημένο μήνυμα. Ε, και έτσι διατηρούμε και το να επιμείνουμε. Θα, ε, τελευταίο σημείο είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών έχει μεγάλη εμπειρία για αυτό το θέμα και είναι μάλιστα το νόημα ε, αυτής της Επιτροπής που έχει άμεση επαφή ε, με τους Ευρωπαίους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν πως εάν η Επιτροπή με αναφορών μπει σε δεύτερο επίπεδο θα είναι κάτι το αρνητικό, ένα αρνητικό μήνυμα. Αντίθετα, θα πρέπει, το, το αντίθετο θα σημαίνει μια ενίσχυση της σχέσης με τους Ευρωπαίους πολίτες. Και υπάρχει και ένα ακόμα επιχείρημα, ότι οι δύο επιτροπές είναι παραπληρωματικές στην εργασία τους. Να μην ξεχνάμε ότι η το νόημα αυτής της πρωτοβουλίας των πολιτών είναι να προωθήσουν πρωτοβουλίες νομοθετικές. Αλλά αυτό που πετύχαμε εμείς ως εμπειρία στην Επιτροπή Αναφορών είναι να φροντίζουμε και να έχουμε αρμοδιότητα και για την εφαρμογή των ε, νομοθετικών κειμένων που υπάρχουν. Δηλαδή δεν εφευρίσκουμε τίποτα, α ε, χρησιμοποιήσουμε και α επωφεληθούμε από την εμπειρία που έχουμε ήδη ισορρεύσει μέσα στο πνεύμα καλή συνεργασία, αγαστή συνεργασία ανάμεσα στι δύο επιτροπέ και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία ανάμεσα στου εισηγητέ και του σχεδόν εισηγητέ των Επιτροπών για να ξεκαθαρίσουμε το ρόλο του καθενό και κυρίω ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε ε, να απευθύνουμε στου Ευρωπαίου πολίτε ω βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μπρόν. Yes, I don't think there's... Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία πιθανότητα ένα εκατομμύριο άτομα από 7 διαφορετικά σε χώρες να προκύψουν, να καταλήξουν σε μια νομοθετική πρόταση κατά το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτό θα συμβεί μόνο αν υπάρχει οργάνωση της κοινή γνώμη και αυτό το περιμένω και το φοβάμαι. Το φοβούνται τα πολιτικά, είτε από τις πολιτικές ομάδες, είτε από τα λόμπι, είτε από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η ιδέα μιας ακρόασης για... είναι ίσως ε, επιφανειακά ενδιαφέρουσα, αλλά σημαίνει διάκριξη μεταξύ αυτών που θα εγκριθούν και που δεν θα εγκριθούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια, ότι είναι συνταγή για την αυτόνομη συμμετοχή. Όχι, πρόκειται για απλά για οργάνωση του κοινού από αυτούς που έχουν ήδη την ε, δύναμη στα χέρια τους και θέλουν απλά δημοκρατική νομιμότητα. Τούτων λεχθέντων υποστήριξα την ιδέα των προτάσεων και τις υπερψήφισα ως τώρα γιατί, γιατί καλύτερο είναι από το τίποτα και γιατί η διαδικασία συλλογής υπογραφών, ακόμα και αν είναι καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως πιστεύω εγώ, θα δώσει στην κοινή γνώμη ένα κίνητρο κινητοποίηση, για να εκφραστεί ίσω με άλλους τρόπου μέσω των εκλογών, μέσω ενός δημοψηφίσματος και γι' αυτό υποστηρίζω την ιδέα της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών και όχι επειδή είμαι αφέλη και πιστεύω ότι θα πετύχουν ποτέ. Κύριε Μποστινάρο, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, θέλω να σας πω εξ αρχής ότι στηρίζω απόλυτα τα όσα υπόθηκαν από όλου του ε, συναδέλφου από την Επιτροπή Αναφορών. Διότι εντό τη Επιτροπή Αναφορά όλε οι πολιτικέ ομάδε μέσω των συντονιστών του και των μελών του στηρίζουν απόλυτα την, ε, την τροπολογία. Πράγμα που δείχνει σαφή ομόφωνη ε, πολιτική στήριξη. Αλλά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για μια εγωιστική προσέγγιση από πλευρά τη Επιτροπή Αναφορών. Είναι το αντίθετο. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε ούτε εξουσίε ούτε να περιορίσουμε τι αρμοδιότητε. Απλώ ε, θέλουμε να κάνουμε μια φιλική ε, ε, έκκληση να σκεφτείτε τη δυνατότητα η Επιτροπή Αναφορών να έχει έναν θεσμικό ρόλο. Εσεί είστε οι πιο καλά εξοπλισμένοι για να ασχοληθείτε με τις πρωτοβουλίες των πολιτών από τη στιγμή που πληρώνται οι προϋποθέσεις. Ταυτόχρονα όμως η Επιτροπή αναφορών όχι μόνο γιατί από κοινού συντάξαμε τις εκθέσεις και ήταν μια μεγάλη επιτυχία όταν ε, διερευνούσαμε μη χαρτογραφημένες περιοχές. Τώρα όμως είναι πολύ σημαντικό να παίξουμε και τον θεσμικό μας ρόλο μαζί σας εξ αρχής γιατί, γιατί αν ε, ληφθεί απόφαση να γίνει η πρωτοβουλία των πολιτών και να ε, εξεταστεί ως ε, ε, αναφορά, να το ξέρουμε και να το κάνουμε αυτό από την αρχή. Επίσης μιλήσατε για την Επιτροπή ΑΦΚΟ και που είναι για μένα σημαντική, αλλά άλλες επιτροπές μπορούν να συμμετέχουν ε, τη στιγμή που η πρωτοβουλία των πολιτών ε, αναφέρεται σε συγκεκριμένους τομείς όπου η δική σας επιτροπή που έχει τον ηγετικό ρόλο και εμείς ως διευτερεύον ε, ρόλος, εκεί λοιπόν να συμμετέχουν αυτές οι επιτροπές ώστε να διερευνώνται συγκεκριμένες, συγκεκριμένοι τομείς όπου είναι σημαντικές οι δικές τους νομοδιότητες. Καλωσορίζω λοιπόν την ε, πρόταση του συναδέλφου Γκερέρο και τις ε, προτάσεις που στήριξαν όλοι οι άλλοι ομιλητές και ελπίζω ότι μετά από αυτή την συνάντηση ανάμεσα σε συντονιστές και οι θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ευέλικτη σοφή λύση που θα είναι ε, ωφέλιμη για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να δείξουμε ότι η δημοκρατία λειτουργεί και ότι τα κενά ανάμεσα στους πολίτες και τα θεσμικά όργανα ε, μειώνεται. Δέχομαι λοιπόν αυτή την ιδέα να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες γιατί δεν έχει να κάνει με τον εγωιστικό ρόλο οποιασδήποτε από τις επιτροπές, αλλά το, με το πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο για την ολοκλήρωση της ζήτησης συνάδελφο Λαμασούρη, θέλω να πω και εγώ κάτι, να προσθέσω κάτι να προσθέσω κάτι για αυτό το θέμα που νομίζω ότι είναι μεγάλη η περιπλοκότητά του από ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Καταρχήν θα τόνιζα τη διαφορά ανάμεσα στην αναφορά και την πρωτοβουλία των πολιτών, που δεν είναι μόνο τυπικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν αφορά μόνο τον αριθμό των υπογραφών και τη δικασία καταγραφής, όχι. Ε, είναι το γεγονός ότι αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών θέλει να συμβάλλει στην εξέλιξη, στην ανάπτυξη των πολιτικών ε, δραστηριοτήτων στην Ένωση, στο σύνολό τη. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για ε, αρμοδιότητες ανάλογες με αυτές που έχουν τα κοινοβούλια και Κομισιόν η ίδια. Πρώτο σημείο. Αυτό πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή η πρωτοβουλία των πολιτών τι θέλει να αλλάξει. Θέλει να αλλάξει κάτι, να πετύχει κάτι και στρέφεται στην Επιτροπή. Δηλαδή ο παραλήπτης είναι η Κομισιόν στην πραγματικότητα, όχι το Κοινοβούλιο. Γιατί λέει η συνθήκη της Λισαβόνας ότι είναι έτοιμα που, στέλνετε, που στην Κομισιόν. Εμείς με τα το 2011 θέλουμε να έρθει εδώ για την Κομισιόν, πρέπει όμως να είναι, μπλέκεται, γιατί αυτή πρέπει να προβεί σε πρωτοβουλία και να λάβει απόφαση. Αυτή είναι μια πολύ βασική διαφορά. Όμως, δεν συμφωνώ, κύριε Λαμασούρ, με το γεγονός ότι η πρωτοβουλία των πολιτών αφορά απαραίτητο μια νομοθετική διαδικασία ή δραστηριότητα. Γιατί η συνθήκη της Λισαβόνα μιλά για νομική πράξη που θεωρείται απαραίτητη για την εφαρμογή των συνθήκων και 188 της συνθήκης λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώ διακρίνει τις, πράξεις, τις νομικές πράξεις μη νομοθετικέ από τι νομοθετικέ. Οπότε θεωρώ πω μπορεί να ζητηθεί και μια γνωμοδότηση, μια σύσταση, μια έρευνα, ένα λευκό βιβλίο Όλε αυτές οι δραστηριότητες που δεν είναι άμεσα νομοθετικές. Δεν το περιορίζω εγώ σε αυτό. Και αυτή είναι μια διάκριση που έχει σημασία. Γιατί, παράδειγμα, όσον αφορά την νομοθετική πράξη, τα επιχειρήματα υπέρ τη επιλογής μιας διαδικασία που θέτει την ακρόαση υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου, γιατί έτσι λέει το άρθρο 211 το 2011, δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε. Θα μπορούσε να γίνει ακρόαση και με την Κομισιόν, που είναι το όργανο που πρέπει να κινηθεί μετά. Άρα λοιπόν η Κομισιόν πρέπει να συμμετέχει από την αρχή και η ιδέα του να συμμετέχει μια αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας, κυρίως όταν ε, πρόκειται για νομοθετική πράξη, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί όπου δεν είναι όμως νομοθετική πράξη, ίσως, ίσως θα πρέπει να δούμε αν υπάρχει αυτή η, πιθανότητα να ανατεθεί αλλού η αρμοδιότητα. Είναι προβληματικό το θέμα, δεν έχω καμιά συνταγή στην τσέπη μου. Μάλιστα συμμερίζομαι την πρόταση που έκανε ο κύριος Λαμασούρα και νομίζω πως είναι δίκαιο να δοθεί και ο λόγος στον κύριο Λαμασούρα για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περίεργος ο σχηματισμός. Πιο πολύ από την Επιτροπή ναι. Αναφορών είναι εδώ από ότι μέλη της δικής μας Επιτροπής. Τέλος πάντων. Και είμαι στο εδόλιο του κατηγορουμένου και στη θέση του εισηγητή, χωρίς να το θέλω. Τέλος πάντων, για να είμαι ειλικρινής. Κοιτάξτε, μπορούμε να τα κάνουμε τώρα, να βρούμε μια λύση. Δεν είναι πρόβλημα. Όλες οι επιτροπές οργανώνουν δύο φορές το μήνα ακρόαση. Ξέρουν να το κάνουν αυτό το πράγμα όλες οι επιτροπές. Δεν είναι ένα θέμα για το οποίο θα κάνουμε και φίλο πόλεμο μεταξύ μας. Τώρα για τη μέθοδο εργασίας. Ο συνάδελφος Ιεύνερ μίλησε για τους τέσσερις ηγητές, ε, τέσσερις άγγελες αποκάλυψης, τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε το θέμα είναι δύο ουσιαστικά ε, κανονισμοί. Εγώ είπα να μην είμαι συγητής, τέλος πάντων. Δεν κάναμε πολλή συζήτηση πριν, θα το κάνουμε τώρα και θα βρούμε λύση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω. Πολλοί από την Επιτροπή Αναφορών, πολλοί συνάδελφοι από την Επιτροπή Αναφορών ανέφεραν την ε, αρμοδιότητα και ίσως και την ε, πρωτοκαθεδρία της Επιτροπής ε, ΑΦΚΟ. Δεν προτείνεται όμως αυτό. Στις τροπολογίες λέγεται ότι η αρμόδια επιτροπή που θα οργανώνει τις ακροάσεις είναι η ΑΦΚΟ. Δεν προτείνεται αυτό. Να ξανάρθουμε στις παρομοίες το ζωικό βασίλειο. Δεν έχει σκύλει αυτό το, σε αυτή τη μάχη το ε, η Επιτροπή ΑΦΚΟ, όπως λένε και οι Άγγλοι σε μια παροιμία. Αυτό που προτείνεται και αυτό που προτείνουμε είναι η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών να αποφασίσει κατά περίπτωση ποια θα είναι η εκάστοτε αρμόδια καθήλυνα επιτροπή. Ο συγκεκριτής περιορίζει ε, στη δυνατότητα να οριστεί μόνο μία επιτροπή ως καθήλαρμο. Θα μπορούσε να είναι πάνω από μία. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχουμε τα άρθρα 50 και 51 που το ορίζουν αυτό, αλλά αφού πρόκειται για νομοθετικό έργο, ε, ξέρουμε τι γίνεται. Πολλέ φορέ όμω έχουμε συνηθίσει να συνεργαζόμαστε για διάφορα θέματα με δύο και τρει επιτροπέ. Παραδείγματο χάρη, διακυβερνητική, διακυβερνητική συγγνώμη, συνεδρίαση σε τρει εβδομάδε πολύ σημαντική με την Επιτροπή ΕΚΟΝ, Αμπλούα και Προπολογισμών. Άρα ξέρουμε να συνεδριάζουμε από κοινού και να οργανώνουμε από κοινού πράγματα. Γίνεται σε τακτά διαστήματα. Το ότι μια στις 10 περιπτώσεις που θα πρόκειται για αρμοδία της Επιτροπής Αναμυντικών Υποθέσεων, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από μια πρωτοβουλία των πολιτών μπορεί να μην είναι πάντα νομοθετικό θέμα που να αφορά κάποια νομική πράξη. Αλλά η ΑΦΚΟ εγώ νομίζω ότι ποτέ σχεδόν δεν θα κριθεί ως καθήλη αρμόδια επιτροπή. Και πρέπει να σας πω το εξής. Ρητά αποκλείει η συνθήκη. Ο Άντρου Ντάφ ε, εξέφρασε και την ε, λύπη του γι' αυτό. Αποκλείει λοιπόν το να αφορά μια πρωτοβουλία την αλλαγή των συνθήκων ή μια σταγματική μεταρρύθμιση. Άρα δεν πρόκειται να δική μας η Επιτροπή Αρμόδια. Η διάσκεψη των πρώτων επιτροπών, κατά περίπτωση παραλαμβάνω, λαμβάνει την απόφαση, εσείς, εμείς τέλο πάντων συμμετέχουμε. Και εγώ διαπιστώνω ότι κάθε φορά που μια επιτροπή, όχι η καθένα αλλά κάποια άλλη επιτροπή ζητά να συμμετάσχει. Να συμμετάσχει στην οργάνωση μια εκδήλωση ή να συντάξει γνωμοδότηση. Η διάσκεψη των πρόεδρων των επιτροπών σπάνια αρνείται. Συνήθω λέει ναι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι συμβατό. με την ε, σύνδεση, τη συστηματική αν θέλετε, αν το ζητήσει βέβαια, της Επιτροπής Αναφορών. Ένα θέμα που θεωρώ σημαντικό από πολιτικής πλευράς είναι το εξής. πρέπει να φάνηκε να είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν διαφορετικέ διαδικασίε. Άλλη διαδικασία ισχύει για τι ευοδοθήσει πρωτοβουλίε των πολιτών και άλλο για τι μη ευοδοθήσει. Αλλιώ δεν έχει καμία ε, σκοπιμότητα και κανένα νόημα να υπάρχει η πρωτοβουλία των πολιτών. Επίση πρέπει να φανεί ότι είναι τελείω διαφορετικό πράγμα από τι αναφορέ οι πρωτοβουλίε των πολιτών, γιατί πάλι δεν θα χρειαζόταν μια τέτοια πρωτοβουλία. Πόσοι πολίτες γνωρίζουν ότι υπάρχει διαδικασία των αναφορών. Mm. Κάποιες χιλιάδες. Πώς γνωρίζουν ότι υπάρχει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητή. Πάλι κάποιες χιλιάδες, ενώ είναι χρήσιμες και οι δύο διαδικασίες. Και η προσφυγή στο Διαμεσολαβητή και η προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών. Εμείς θέλουμε να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Προστιθέμενη αξία που θα δείξει ότι αν οι Ευρωπαίοι πολίτες οργανωθούν και αν οργανωθούν και πέραν των συνόρων, διασυνοριακά, γύρω από ένα θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση, μπορούν να έχουν πολιτική εξουσία ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ισοδύναμε με αυτή του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το θέμα. Τη στιγμή λοιπόν που ο κανονισμός προβλέπει δημοσιακρόαση, αυτή η δημοσιακρόαση θα πρέπει να οργανωθεί κατά τρόπο εντελώ διαφορετικό από αυτόν τον οποίο οργανώνεται η διαδικασία εξέταση αναφορών. Θα μπορούσε αυτό να γίνει με τη συνδρομή τη Επιτροπή Αναφορών. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι θα έχει το μονοπόλιο η Επιτροπή Αναφορών, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι σαφέ ότι χρειάζεται μια διαδικασία η οποία θα παρέχει όλα τα εχέγγυα και θα έλεγα και να δίνει και μια επισημότητα, αλλά να είναι διαφορετική από την τακτική, την κανονική διαδικασία που ακολουθεί η Επιτροπή Αναφορών. Και το λέω και το παραλαμβάνω. Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να υποβαθμίσω τον πολύ σημαντικό ρόλο τη Επιτροπή Αναφορών. Δεν θα είχαμε καμία επαφή με τον πολίτη αν δεν υπήρχε αυτή η Επιτροπή. Αλλά από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, τίνω να διατυπώσω δύο προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, σε ό,τι αφορά μέθοδο, Νομίζω και θα προσπαθήσω να επηρεάσω ε, την εισηγήτρια για να την πείσω και δεν νομίζω να δυσκολευτώ ιδιαίτερα. Θα συναντηθούμε οι λίγοι αυτοί συνάδελφοι των δύο επιτροπών που ενδιαφερόμαστε για το θέμα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και σε συνάρτηση με την έκβαση αυτών των συνομιλιών θα σας πρότεινα, αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, πριν, θέσουμε σε ψηφοφορία αυτή την έκθεση στην Επιτροπή ΑΦΚΟ, σε μια προσεχή συνεδρίαση της διάσκεψης των πρώτων των Επιτροπών, να θέσουμε το θέμα για να δούμε ποια είναι η άποψη των άλλων Πρόεδρων των Επιτροπών. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και στην Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών να επιχειρηματολογήσει υπέρ ε, τη ε, πρότασή τη. επειδή για αυτή τη νέα διαδικασία η λύση που θα επιλεγεί θα εξαρτηθεί από τη φιλοσοφία που θα ακολουθήσουν οι αρχές του Κοινοβουλίου για τον επιμερισμό των καθηκόντων μεταξύ των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών και επειδή η δημιουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών και ο επιμερισμός των αρμοδιοτήτων εξαρτάται από απόφαση που λαμβάνει η Ολομέλεια βάση προτάσεως στη διάσκεψη των Επιτροπών, νομίζω ότι είναι ένα θέμα που καλό θα ήταν να ε, συζητηθεί, να γίνει μια παρουσίαση και συζήτηση στην ε, διάσκεψη των πρώτων των Επιτροπών. Και μετά θα ψηφίσουμε και πιστεύω να βρει ευρεία υποστήριξη το κείμενο το οποίο θα συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαμασούρ. Νομίζω πως μπορούμε να κλείσουμε αυτή την σημαντική και επικοδομητική συνάντηση και έτσι με την οποία εμπλουτίσαμε τη σκέψη μας. Σας ευχαριστώ. Τέλος της συνεδρίας. ευχαριστώ τους συναδέλφους της Επιτροπής Αναφορών.